Buenos días. Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ, καθίστε να ξεκινήσουμε. Έχει έρθει ήδη η Επίτροπος η κυρία Γιούροβα. Ξέρετε πως είναι η αρμόδια για την δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ισότητα των φίλων; Η δικαιοσύνη είναι βασικό ζήτημα για την Επιτροπή μας. Όπως είχα την ευκαιρία να ε, σχολιάσω μαζί σας, είχαμε μια πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στην αρχή της Φιλανδικής Προεδρίας. Είχε έρθει εκεί πέρα η κυρία Γιούροβα και ζήτησε ε, δικαστική συνεργασία στα ποινικά ζητήματα και όχι μόνο και για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, προστασίας ε, δεδομένων για ζητήματα κράτους δικαίου σύμφωνα με το μηχανισμό που υιοθετήσαμε στο τέλος της ε, προηγούμενης ε, θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίω όσον αφορά την οδηγία περί μεταχείρισης ε, που εκκρεμεί 11 χρόνια ήδη. Και αρκετοί από εσά θέσατε το θέμα στον ε, κύριο Τζούλιαν Κίνγκ, τον Επίτροπο. Οπωσδήποτε η κυρία Γιουροβά θα μας αναπτύξει τις απόψεις της, όπως έκανε και στην ε, προηγούμενη εντολή, στην προηγούμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την καλωσορίζουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε με ερωτήσεις, ε, δύο λεπτά ο καθένας από τους συντονιστές και μετά θα περάσουμε και στους υπόλοιπους βουλευτές. Αλλά όσοι ενδιαφέρεστε να μιλήσετε στο δεύτερο γύρο και όλοι οι βουλευτές ε, μπορούν, ε, παρακαλώ σηκώστε την κάρτα σας για να μιλήσετε στον δεύτερο γύρο. Κυρία Γιώροβα, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και για το ότι είστε σε αυτήν την σημαντική επιτροπή. Τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν στην προηγούμενη θητεία είναι πολύ σημαντικά για την σημερινή κοινωνία και ο κύριος Πρόεδρος ήδη ανέφερε τα θέματα αυτά ασφάλεια κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και καταπολέμηση των διακρίσεων. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, βουλευτές ε, που ε, επέλεξαν αυτήν την επιτροπή, ειδικά σε μια στιγμή στην οποία ο ρατσισμός και η ξενοφοβία αυξάνεται στην Ευρώπη. Πέρα το ότι βεβαίω πλησιάζουμε στο τέλος της θητείας της Κομισιόν, εργαζόμαστε σε κάποια πολύ βασικά ζητήματα και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις και να ακούσω τις απόψεις σας. Έχουμε διάφορα θέματα και δεν έχουμε αρκετό χρόνο να τα καλύψουμε. Ευχαριστώ βεβαίω να σας πω όλα όσα ξέρω. Έπρεπε όμως να γίνει μια επιλογή ε, κάποιων ε, θεμάτων για συζήτηση σήμερα. Οπότε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην ανακοίνωση για το καρτσοκέο το πακέτο εκθέσεων για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, και η ταυτοποίηση τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου επίσης θα αναφερθώ στην ανακοίνωσή μας για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αλλά και την ασπίδα προσωπικών στοιχείων που έχουμε με τις ΕΠΑ και τον κανονισμό περί αποδεκτικών στοιχείων και θα σας ενημερώσω με το πώς προετοιμάζεται να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελπίζουμε του χρόνου. Θα ξεκινήσω με το κράτος ε, δικαίου που ήταν σαφώς ένα από τα βασικά ζητήματα στις ε, συζητήσεις που είχαν οι πολιτικές σας ομάδες με την ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Μετά από διαβουλεύσεις και κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Κομισιόν προτείνει τις εξής δέσμες δράσεις για να ενισχυθεί το κράτος δικαίου. Ε, μια ετήσια έκθεση κρατου δικαίου που θα καλύπτει όλα τα κρατη με ρόλο προληπτικό. Έτσι θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις σε Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Μια διαδικασία ε, παραβασιών που θα είναι πιο στρατηγική και θα βασίζεται στην ομολογία του κρατζοκαίου. Η ενίσχυση της κουλτούρας κράτους δικαίου στο κοινό. Αυτό σημαίνει να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες χρηματοδότησης ε, για την κοινωνία των πολιτών για να προωθήσουμε το κράτος δικαίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα μπορούσαν επίσης να αναπτύξουν συγκεκριμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία στα ζητήματα αυτά, στα οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει και η Κομισιόν επιπλέον. Η Κομισιόν θεωρεί ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει στην διαδικασία του άρθρου 7 ξεκάθαρους και σταθερούς κανόνες ε, και εμπλοκή του Κοινοβουλίου στην περίπτωση που έχει ξεκινήσει τη διαδικασία, όπως είχε ήδη γίνει. Τέλος, το σχέδιο κανονισμού για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης σε περίπτωση ελλείψης στο κράτο δικαίου στα κράτη-μέλη θα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, όπως ακούσαμε από την Φιλανδική Προεδρία, ε, σκοπεύουν να το προωθήσουν. Η Κομισιόν συνεχίζει το έργο της στην καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος μετά τα πολλά σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια. Χτες εγκρίναμε μία σειρά σημαντικών εκθέσεων για να εξετάσουμε τις υπάρχουσες ανάγκες και το τι πρέπει να βελτιωθεί. Υπάρχουν ε, πάρα πολλά πράγματα στην έκθεση. Σημαντικά θα αναφερθώ μόνο σε μερικά κυρία συμπεράσματα. Η συμμόρφωση με τους κανόνες ε, είναι ανεπαρκής και η εποπτεία των ε, αρμόδιων αρχών αδύναμη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Επλέον υπάρχουν συγκεκριμένοι κίνδυνοι όπως οι ανώνυμες συναλλαγές, έλλειψη διαφάνειας ε, πραγματικού ιδιοκτήτη και νέες τάσεις όπως ε, η εικονική χρήση. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά με διάφορους τρόπους μεταξύ των οποίων η τέταρτη και πέμπτη οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος, η οδηγία περί χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, η αναθεωρημένη οδηγία περί οικονομικών πληροφοριών και η συνεργασία των εποπτικών αρχών. Η Κομισιόν παίρνει πολύ σοβαρά τον ρόλο της ως θεματοφύλακας των συνδικών και έχει αρχίσει διαδικασίες κατά όλων των κρατών μελών λόγω της πλημελού εφαρμογής ε, της ε, τέταρτης οδηγίας πολέμηση ξυπλήματος ε, χρήματος. Πολλά έχουν γίνει λοιπόν, αλλά η δουλειά μας ακόμα δεν έχει τελειώσει, όπως αναφέρει και η κύρια Ωσουλα Φαντερ πρέπει να κλείσουν τα παραθυράκια. Το σχετικό πακέτο το οποίο εγκρίθηκε χτες μας δίνει μια βάση για την περαιτέρω συζήτηση ειδικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παραδείγματος χάρη περαιτέρω εναρμόνιση και ένας κανονισμός ο οποίος θα ισχύει απευθείας και θα αφορά το ξέπλυμα χρήματος και θα αναθέτει τα καθήκοντα αυτά σε έναν φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, με βάση τα όσα πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για να διασφαλιστεί συντονισμός μεταξύ των μονάδων χρηματοπιστωτικών πληροφοριών στα κράτη-μέλη. Για την εξωτερική ε, πλευρά, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται την μεθοδολογία για τις χώρες υψηλού κινδύνου από την σκοπιά ξεπλήματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εδώ ακολουθούμε τις ε, αντιρρήσεις ε, του Συμβουλίου. Πρόκειται όμως για μια νομική υποχρέωση και κοινή ευθύνη και των τριών θεσμικών οργάνων. Μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαρτίου εργαζόμαστε προς μια διαδικασία με διαφάνεια με σαφή κριτήρια για τις χώρες οι οποίες θέλουν να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για να μην μπουν στον κατάλογο. Χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για να διασφαλίσουμε το ότι το Συμβούλιο θα αποδεχτεί την μεθοδολογία και θα είμαστε σε επαφή με το Κοινοβούλιο και με τους συναδέλφους σας στην Επιτροπή Οικονομικών και θα θέσω το ζήτημα και με τους Υπουργούς ε, Οικονομικών Συμβουλίου Κοφήν τον Οκτώβριο. Χρειάζεται να ανοίξουμε τον δρόμο ε, στο ζήτημα αυτό. Παράλληλα, έχουμε εντείνει τις επαφές μας με τις ε, τρίτες χώρες και ενισχύουμε τον ρόλο της Κομισιόν στην ε, ομάδα δράσης, η οποία προσφάτως έβαλε και τον Καναδά στις χώρες υψηλού κινδύνου και επιβεβαιώνει έτσι την αξιολόγηση της Κομισιόν που έγινε τον Φεβρουάριο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις διαφορές μεταξύ του καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας δράσης. Αυτά για το ξέπλυμα χρήματος. Να επιτρέψατε μου τώρα να αναφερθώ σε ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της Επιτροπής σας, ε, την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Σώμα των Επιτρόπων χτες ενέκρινε μια αξιολόγηση της λειτουργίας ε, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ε, τα συμπεράσματά μας είναι ότι λειτουργεί καλά. Βλέπουμε ενιαία εφαρμογή στα κράτη-μέλη, ισχυρότερη επιβολή και οι ε, επιχειρήσεις το θεωρούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες πτυχές βεβαίως, κάποια κράτη-μέλη πρέπει ακόμα να προσαρμόσουν την ε, νομοθεσία τους και να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή κουλτούρα ιδιωτικότητας. Πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αντιληφθούν καλύτερα το τι πρέπει να κάνουν. Και βεβαίως το κοινό γνωρίζει τον κανονισμό και αυτό μας ικανοποιεί, αλλά θα μπορούσε ο κόσμος να δρά πιο προληπτικά αποτελεί πλέον ένα σημείο αναφοράς ενός ε, υψηλού επίπεδου Προστασία σε άλλες χώρες, στην Ασία, τη Λατινική Αμερική, την Αφρική, αλλάζουν την ε, νομοθεσία τους ε, και έχουν ως σημείο αναφορά στον κανονισμό μας. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία θέτει τους κανόνες. Επίσης, και άλλες χώρες θέλουν να αντιγράψουν την συμφωνία μας με την Ιαπωνία, όπως η Νότια Κορέα. Είχα πάει στην Αργεντινή πριν από 15 μέρες. Η Χιλή επίσης συντάσσει τον πρώτο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο οποίος είναι εμπνευσμένο από τον δικό μας κανονισμό. Η Αργεντινή επίσης αλλάζει τον νόμο της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πλαίσιο των εμπορικών συμφωνιών μας με τις δύο χώρες αυτές. Ακόμα και στη ΣΥΠΑ, Ε, συζητιέται η αλλαγή της ε, νομοθεσίας τους. Το τελευταίο ε, πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που, δολαρίων με που επέβαλαν οι Αμερικανικές αρχές στο Facebook αποτελεί μια ένδειξη. Θα πρέπει ε, να δούμε βεβαίως ε, τι ακριβώς ε, σημαίνει. Και αναφέρεται το πρόστιμο αυτό στην υπόθεση της Cambridge Analytica. Και έρχομαι τώρα στην ασπίδα προσωπικών δεδομένων. Επίσης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην ευρωπαϊκή πλευρά και κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να εγγυηθούμε την προστασία της ιδιωτικότητας στο αμερικανικό έδαφος. Ως απόδειξη αυτού, πάνω από 4.700 εταιρείες έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο πλαίσιο αυτό. Παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή του και η πίεση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι πάρα πολύ χρήσιμη για να προχωρήσουν τα πράγματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ορίστηκε η μόνιμη επίτροπος όπως ε, επίσης και το Εποπτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και μία προσέγγιση από το Υπουργείο Εμπορίου για να ελέγχει τις συμφωνίες μεταξύ εταιριών. Θα τα δούμε αυτά στο τέλος της ετήσιας ε, εξέτασης μου που θα γίνει πριν το τέλος της ε, θητείας μου. Οπότε φαίνεται ε, πηγαίνουμε προς τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η ασπίδα αυτή η ιδιωτικότητα αφορά την μεταφορά προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εμπορικών σχέσεων, αλλά υπάρχει διατλαντική συνεργασία και στον τομέα των διοκτικών αρχών. Όπως ξέρετε, τα δεδομένα ταξιδεύουν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό βεβαίως αποτελεί ένα πρόβλημα για τους εισαγγελείς και το σύστημα α, της δικαιοσύνης που έχει κάποια δυσκολία στο να έχει πρόσβαση στα ηλεκτρονικά δεδομένα. Και η μορφή αυτή των στοιχείων πλέον χρειάζεται σε ένα 85% όλων των ποινικών ερευνών. Δηλαδή ουσιαστικά σε κάθε έρευνα πλέον ε, χρειάζονται ηλεκτρονικά δεδομένα. Η διαδικασία απόκτησής τους είναι πάρα πολύ ε, αργή και αυτό εμποδίζει τις έρευνες, κάτι το οποίο τελικά σημαίνει ατιμορρησία και επηρεάζει την εμπιστοσύνη στο σύστημα της δικαιοσύνης από την πλευρά των θυμάτων. Γι' αυτό έχουμε αυτό το πακέτο ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Έτσι θα μπορούν ε, οι πάροχοι γρήγορα να δίνουν αυτά τα δεδομένα, σεβόμενοι πάντα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Συμβούλιο ενέκρινε μια γενική προσέγγιση στα τέλη του προηγούμενου έτου. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε μια θέση έτσι ώστε οι διοργανικέ διαπραγματεύσει να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν. Η Κομισιόν είναι στην διάθεσή σα για να στηρίξει αυτήν την διαδικασία. Έρχομαι τώρα στην διεθνή διάσταση το Συμβούλιο έδωσε μια εντολή στην Κομισιόν στις 6 Ιουνίου για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ηλεκτρονικά αποδεκτικά στοιχεία και να συνυπογράψει τα τέσσερα σχετικά πρωτόκολλα της Βουδαπέστης. Έχουμε ένα συμφέρον για να περιορίσουμε την ε, εξοδαφική ισχύ των Αμερικανικών νόμων. Σκοπεύουμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ μόνο όταν συμφωνήσουμε εσωτερικά στους κανόνες. Οπότε πριν συμφωνήσουμε στους κανόνες για τα ηλεκτρονικά αποδεκτικά στοιχεία, λογικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η προσέγγιση μας ε, διαφέρει από την Αμερικανική νομοθεσία. Εμείς θέλουμε μια νομοθεσία η οποία θα είναι σωστή για την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να διασφαλίσουμε η συμμεταχείριση όλων των ατόμων. Είναι προς το συμφέρον μας η να συνάψουν ε, διμερείς συμφωνίες με κάποιε φορέ όχι όμως με κράτη-μέλη, γιατί στην περίπτωση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει την δυνατότητα εποπτείας. Οπότε θα σε ενημερώσω τους επόμενους μήνες για όλες τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι τα διαδικαστικά δικαιώματα και οι δικλείδε ασφαλείας θα πρέπει να περιληφθούν στην τελική συμφωνία. Τέλο, στον τομέα του ποινικού δικαίου πάντα σημειώνουμε πρόοδο προς την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής εισαγγελία που θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί στο τέλος του 2020. Η Κομισιόν έχει ξεκινήσει την απαραίτητη προεργασία αλλά είναι πλέον επίγον Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που θα παίξει και κέριο ρόλο στη λειτουργία της υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, στην Επιτροπή σας ασχοληθείτε και με θέματα τα οποία σχετίζονται με τα πιο σημαντικά και επίγοντα ε, ζητήματα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η προστασία των εθνοτικών μηνοτήτων ε, και ούτω καθεξής. Στο περιορισμένο χρόνο που έχουμε στη διαθεσή μας δεν μπορώ σήμερα να τα συζητήσω όλα αυτά, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστώ ε, <clears throat> ακούραστα για όλα αυτά τα ζητήματα μέχρι το τέλος της θητείας μου. Επιτρέψατε μου να αναφέρω μια σημαντική νομοθεσία όπου πιστεύω ότι έχουμε θετικές εξελίξεις. Η Φιλανδική Προεδρία θα αφιερώσει κομμάτι του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ του Οκτωβρίου όσον αφορά την οδηγία που, στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Πρόεδρος όταν μιλούσε για 11 χρόνια εκκρεμότητας εκεί σε αυτό, το, σε αυτό το τομέα όπου Χρειάζεται όμως ομοφωνία στο Συμβουλίο και είμαι ευγνώμων στη Φιλανδική Προεδρία που θέλει να το φέρει τον Οκτώβριο στο Συμβούλιο γιατί πρέπει να αρχίσει και πάλι αυτή η συζήτηση και να προσπαθήσουμε ξανά και ξανά εκεί. Ελπίζω πως αυτή η συζήτηση τον Οκτώβριο θα ε, ε, <clears throat> οδηγήσει σε μια πολιτική εξολόγηση που θα ανοίξει το δρόμο για να μπορέσει να κινηθεί το Συμβούλιο και Απολύτως υποστηρίζω την ε, κίνηση αυτή. Αξιότιμη κύριε Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ πολύ ε, για την προσοχή σας και προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Εσείς διευρύνατε το πεδίο των ε, προβληματισμών που εγώ αρχικά ανέφερα και συμπεριλάβατε εκεί και την προβληματική υπερατλαντική διάσταση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ όσον αφορά την ε, νομοθετική διαδικασία ε, ε, εφόσον αφορά τα στάνταρ προς προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων για ιδιωτικότητα, για προστασία προσωπικών δεδομένων και επικοινωνιών και βέβαια για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Όπου υπάρχει μια μεγάλη και διελκυστίνεται ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τούτων λεχθέντων, για το πρόβλημα της οριζόντιας οδηγίας για την ίση μεταχείριση και της, ε, των μη διακρίσεων σημαίνει ε, αυτό, απαιτεί μάλλον πρωτοβουλία. Είναι πολύ δυσλειτουργικό αυτό. Ακούσαμε την ε, πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Μαντερλάιεν να προβληματίζεται και εκείνη με τον κανόνα της ομοφωνίας, να μπορέσουμε να βρούμε πασαρέλες σε, με κάθε δυνατό τρόπο και τώρα πρέπει να ακούσουμε τους συντονιστές μας ώστε ε, να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο και στους υπόλοιπους συναδέλφους που θέλουν να παρέμβουν. Να είστε σύντομοι παρακαλώ. Ξεκινάμε με το ΕΛΚΑ. Ο συντονιστής η συντονίστρια Μετσόλα και Ελένα δεν είναι εδώ, αλλά θα εκπροσωπηθούν από τον κύριο Πίτερ σε αυτό το πρώτο γύρο. Σωστά, μάλιστα, σωστά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, ευχαριστώ και σας συγχαίρω για όλη την ε, εργασία σας τα τελευταία χρόνια. Αναφέρατε πολλά ζητήματα βέβαια. Θα κάνω μία σύντομη επισκόπηση και κάποιες ερωτήσεις καταρχάς για την αξιολόγηση του GDPR. Το αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, η ερώτησή μου σε αυτό το τομέα είναι τώρα ποια ε, πού βρίσκεται η συζήτηση όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα γιατί υπάρχει εκεί εξέλιξη μάλλον εάν υπάρχει εξέλιξη και αν πρόκειται να υπάρξει ειδική διάταξη για τον ιδιωτικό τομέα. Έπειτα, για τα τέλη του 2020 είπατε για την ασφαλή ε, ε, ε, για το Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Είναι όμως ρεαλιστικό αυτό. Ε, αυτό ο χρονικός ορίζοντας. Το άλλο μου ερώτημα είναι για το ε, ε, κοινή παροχή στοιχείων όταν πρόκειται για συγκρισιμότητα και ανταλλαγή στοιχείων και δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό να δράσουμε σε αυτό το τομέα. Αν δούμε το B2B data sharing και όταν βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναφέρατε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα των δεδομένων και η τελευταία μου ερώτηση είναι πολύ σημαντική και αφορά το πρόβλημα των ανώνυμων δεδομένων. Αναφέρατε και εσείς αυτό το στοιχείο και γνωρίζετε ότι την Τρίτη Έγινε μια πολύ, παρουσιάστηκε μια πολύ σημαντική έκθεση από συναδέλφους στο Λονδίνο και του Πανεπιστημίου της ε, Λουβέν που δημοσίευσαν ε, την ε, μια έκθεση για τις διαδικτυακές επικοινωνίες. Αυτή η έκθεση λέει ότι μέσω των επικοινωνιών τους οι άνθρωποι μπορούν να εντοπιστούν και να αναγνωριστούν. Είναι πολύ σημαντική η μελέτη, αλλά είναι και πολύ σημαντικό το μήνυμα που προκύπτει από εκεί, ότι δηλαδή έχουμε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Πώς προτίθεστε να παρακολουθήσετε αυτή την αυτή την υπόθεση και τις επιπτώσεις της και πώς μπορούμε να χειριστούμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα τώρα η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να θέσω μια ερώτηση, γιατί φαίνεται ότι ένα και περισσότερο στα κράτη-μέλη μας, κάποια κράτη-μέλη, κάποιες ομάδες πολιτών επηρεάζονται όλο ένα και περισσότερο από ε, ε, το λόγο μίσους και διακρίσεις και κάποιες φορές έχουμε και βίες επιθέσεις. Το είδαμε ας πούμε στην Πολωνία κατά ε, ανθρώπων της ομάδας LGBTI. Ε, η Κομισιόν αναλαμβάνει πιο σοβαρά τις ευθύνες της. Θα πρέπει να το κάνει αυτό για την καταπολέμηση αυτών των ε, δράσεων, αλλά να δραστηριοποιηθεί κιόλα για την καταπολέμηση. Στον τομέα της προστασίας των δεδομένων θέλω να θέσω κάποιες ερωτήσεις. Έγινε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να δούμε πώς ο συνδυασμός διαφόρων βάσεων δεδομένων, επί των οποίων αποφασίσαμε τα τελευταία χρόνια, επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Υπάρχουν ήδη κάποια αποτελέσματα γι' αυτό. Παρόμοια ερώτηση αφορά την οδηγία περί αστυνομίας. Μετά την GDPR ακολούθησε αυτή. Και εδώ υπάρχουν κάποιες επιπλέον, κάποιοι πλέον κανόνες και διασφαλιστικές δικλείδες. Μπορείτε να μας πείτε ε, λίγο πού βρισκόμαστε και αν μπορούμε να έχουμε μια έκθεση για αυτό το θέμα. Άλλη μου ερώτηση αφορά το θέμα της ιδιωτικότητας, <coughs> έχουμε νέα μέλη εδώ και είδα ότι ο αριθμός των εταιριών μετά από αυτού, που, ακολουθούν αυτούς τους κανόνες έχουν αυξηθεί. Εσείς μπορείτε να εξηγείτε με ποιο τρόπο το ελέγχουμε, το πότε αυτές οι εταιρείε που έχουν συνυπογράψει αυτούς τους κανόνες ε, αν πραγματικά ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που αφορούν την ασπίδα ιδιωτικότητα σε συνεργασία με τη ΣΥΠΑ και πώς λειτουργεί αυτό. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά το άρθρο 7. Είπατε ότι μπορεί να χρειαστούμε πιο σαφείς κανόνες για το πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, ώστε να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε αποτελέσματα. Η εντύπωσή μου είναι πως ίσως το πρόβλημα να μην είναι οι σαφέστεροι κανόνες, αλλά η πολιτική βούληση. Ωστόσο, η Κομισιόν έχει ήδη κάποια ιδέα για το ποιοι κανόνες θα είναι αυτοί και τι μορφή θα έχουν. Ευχαριστώ. Ιντεβέλντ, εξ ονόματος του Ρινιού. Μάλιστα σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Με χαρά σας είδαμε σήμερα εδώ. Αναφερθήκατε σε πολλά ζητήματα τα οποία θα ανατρέξω σύντομα. Με χαρά ακούσαμε ότι εξετάζεται έναν κανονισμό για την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο και την εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί το είπαμε και χτε ότι η επιβολή είναι ε, λατωματική, ελλειπή. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων που ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Με την, για την ε, ευρωπαϊκή λοιπόν ε, ε, νομοθεσία. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την αδύναμη πρόταση που προέτεινε ο συνάδελφός σας Τίμερμανς, γιατί το πεδίο εφαρμογή είναι στενό, αφήνονται εκτός θεμελιώδη δικαιώματα και η δημοκρατία εστιάζει αποκλειστικά σε κάποια θέματα. Δεν υπάρχουν συστάσεις για μεμονωμένες χώρες, ούτε προτάσεις για ανεξάρτητου συμπειρογνώμονες. Οπότε εμεί θα υποβάλλουμε ε, τροπολογίες. Ε, Τώρα, καράτος δικαίου. Μιλήσατε για την ιδιωτική επιβολή. Ε, αυτό είναι τμήμα του κράτου δικαίου. Δηλαδή, οι πολίτε ΜΚΙΟ, αυτές μπορεί, αυτοί να, χρειαστεί να βρεθούν αντιμέτωπες ε, και μάλιστα, όπω γνωρίζετε, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ε, ταμείου ε, ρύθμισης διαφορών. Παρά το ότι τα, τις δικές μας εκκλήσεις ε, και ε, την πίεση που έχουμε ασκήσει, τελικά εσείς δεν το χρησιμοποιείτε όπως θα έπρεπε. Πρέπει να γίνει αυτό πραγματικά ένα ταμείο το οποίο θα ενισχύει τους πολίτες που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Τώρα, στη, όσον αφορά τη σχέση μεταξύ ΕΠΑ ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε λίγο υποτακτικοί των ΕΠΑ. ΕΕ. Δεν έχουμε σταθεί στο ύψος μας. Το διαπραγματευτική εντολή θα πρέπει να δημοσιευθεί κατά τη γνώμη μου. Τους άλλους είναι τα δικά μας στοιχεία περί των οποίων πρόκειται. Η εντολή για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με το, Συμβου... Συμβούλιο ε, να δημοσιευθεί. Και τέλος να πω εδώ στους συναδέλφους ότι όταν θα, περάσει, θα έρθει η τελευταία συμφωνία θα πρέπει να υποβληθεί στο ECJ πριν ε, για γνωμοδότηση πριν εμείς να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ευχαριστώ. Είμαστε συνσυντονίστες. Ναι, εντάξει, το συγγνώμη γιατί θα σα ε, δυσχεράνουμε λίγο το έργο σα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας, κύριε Επίτροπε, και όπως είπατε, έχουμε πολλά να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω, γιατί ακόμα και αν μπορεί αυτά να φαίνονται δύσκολα και αντιφατικά, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να κάνετε πίσω. Θα πρέπει να πάμε πιο πέρα από τα όσα έγιναν στην τελευταία θητεία. Να πω δύο πράγματα για τα όσα εσείς αναφέρατε για το μηχανισμό κράτους δικαίου, θα ήθελα να στηρίξω το αίτημα ότι η ανακοίνωση της Κομισιόν που μόλις δημοσιεύθηκε δεν προχωρά αρκετά όσον αφορά τους ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες αλλά και το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πιστεύω θα πρέπει να ανοίξουμε συζήτηση εδώ. Και μια ερώτηση, γιατί αναφέρατε το μέσο έλλειψης κράτους δικαίου για τον προπολογισμό. Πώς θα συνδεθεί αυτό με όλα αυτά, γιατί για μα θα έπρεπε να υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα ε, στις παραβιάσεις κρατός δικαίου και θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη και το Ταμείο αυτού. Ελπίζω ότι η Κομισιόν λοιπόν θα, θα το στηρίξει αυτό. Νομίζω πως είναι πραγματικά κρίμα μετά από 11 χρόνια ως Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορούμε να προχωρήσουμε Ε, ε, για την καταπολέμηση ε, επίσης των διακρίσεων θα πρέπει να πιέσουμε στην επόμενη θητεία να δημιουργηθεί μια στρατηγική για τους LGBTI. Και η τελευταία μου παρατήρηση, είδαμε κάποιες θετικές ενέργειες στο πρόγραμμα της ε, ψήφιας ε, Προέδρου, δηλαδή για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και μια οδηγία για τη βία, ε, την έμφυλη βία. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το κατά πόσο είστε έτοιμοι να κινηθείτε για αυτά τα θέματα, γιατί πιστεύουμε εμείς πως είναι πολύ σημαντικά. ID, κυρία Ταρντίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ. Πολλές, πολλά τα σημεία που αναφέρατε στην εισήγησή σας, εγώ θα σας επικεντρωθώ στην δικαιοσύνη. Την περασμένη Απρίλη υποβλήθηκε το πλαίσιο αξιολόγησης της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολόγηση των δικαστικών συστημάτων και της εφαρμογής της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη σύγκριση προκύπτει σαφώς πως υπάρχουν προβλήματα διάρκειας των διαδικασίων ε, διαδικασιών που κάποιες φορές είναι πολύ μακρές σε κάποια κράτη και προβλήματα με την ε, εισαγγελία. Αντίληψη από πλευράς του κοινού της ανεξαρτησίας ε, ε, του δικαστικού σώματος έχει μειωθεί κατά τα τρία πέμπτη σχεδόν σε όλα τα κρατη Και αυτό είναι δύο πέμπτα στα, στα κρατη Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό όσον αφορά το κράτος δικαίου. Εσείς πώς κρίνετε αυτά τα αποτελέσματα, ποια είναι τα επόμενα βήματα για τις συστάσεις της Κομισιόν και ποιες είναι οι προτεραιότητες προτεραιότητε επί των οποίων θεωρείται ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί ο επόμενο επίτροπο ώστε να επιτύχει συνεργασία με τα κράτη-μέλη και του στόχου που εμεί θέλουμε για του συμπολίτε μα. που περιμένουν πάρα πολύ χρόνο πριν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ποκατσίνη, ECR. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε, κύριε ε, Επίτροπε Γιούροβα. Ευχαριστώ για την εισήγηση. Ε, δεν μπορώ παρά να παρατηρήσω ότι παρότι ε, το χρονικό διάστημα ήταν ε, ευρύ και μακρύ, ε, τελικά η συζήτηση για το κράτος δικαίου, για το άρθρο 7, σκοντάφτει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Στο Ελσίνκι παρατήρησα πως είστε ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με την, το κράτος δικαίου, ωστόσο παρατήρησα πως και εσείς οι ίδια επανειλημμένα αναφερθήκατε σε αυτήν την ε, το περιορισμένο ε, φάσμα αυτής της ε, διάταξης. Αυτό ακριβώς είναι που χρησιμοποιήθηκε για να περιορίσει αυτό το κράτος δικαίωμα. Μα τι έχετε εσείς, έχετε έναν πίνακα πάνω στον οποίο βάζετε από τη μια τους καλούς και από την άλλη τους κακούς και έπειτα ε, υπάρχει ένα είδος ερμηνείας αστυνομικού τύπου όσον αφορά το κράτος δικαίου. Εγώ θα ήθελα μόνο να σας σημειώσω ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει μέσο κυρίως κατά των μειονοτήτων. Και αυτή που είναι αυτή τη στιγμή η πολιτική μειονότητα, ακόμα και εδώ μέσα, σε αυτό την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει πλειοψηφία. Γι' αυτό και επιστήνω ιδιαίτερο στην προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. Γκουε τώρα, δεν βλέπω την Κορνίλια Ένστ. Ο κύριος Πελετ, η κυρία Πελετχέ, η Μαντάμ Πελετιέ, κυρία Πελετιέ. σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την εισήγησή σα. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σα στο δικαίωμα Άμυνα, γιατί υπάρχουν νέα μέσα δικαστική συνεργασία και εμεί ε, προβληματιζόμαστε κατά πόσο αυτά τα δικαιώματα τηρούνται και πόσο είναι εγγυημένα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οθετήσει έξι οδηγίε για τα δικαιώματα στην υπεράσπιση ε, ε, <laughs> Και οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Μπορείτε σήμερα να μας πείτε ποια είναι τα αποτελέσματα που έχετε. Αν έχετε, υπάρχουν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, υπάρχουν ελλείψεις, κενά. Και έπειτα, μήπως έχετε και μια ημερομηνία για την πρώτη σας αναφορά. Και τι θα συστήσετε στον επόμενο επίτροπο ή την επόμενη επίτροπο. Επιστρέφουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 10 λεπτά για να μπορέσετε να απαντήσετε στον πρώτο αυτό γύρο ερωτήσεων των συντονιστών και μετά θα προχωρήσουμε σε επόμενο γύρο, γιατί βέβαια είναι μακροσκελής ο κατάλογος με τα ονόματα των μελών μας που επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις. Σας παρακαλώ λοιπόν, κάντε προσπάθεια να απαντήσετε. Ε, Βεβαίω είναι, θα είναι ε, ε, δύσκολο έργο. Ναι. Όσο περισσότερο είμαστε στην πολιτική, τόσο πιο πολύ δυσκολευόμαστε να τα λέμε σύντομα. Θα προσπαθήσω όμως. Πρώτη ερώτηση. Πέτερς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του GDPR. Νομίζω ότι ε, είναι νομοθέτημα του ψηφιακού τομέα και όχι του ιδιωτικού δικαίου. Όμως, το δήλωσε ήδη η υποψήφια πρόεδρος της ε, Κομισιόν αυτή, το ερώτημα του Άμλετ να νομοθετήσουμε ή να μην νομοθετήσουμε, να ρυθμίσουμε νομοθετικά ή να μην ρυθμίσουμε νομοθετικά. Πάντως, υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν βέβαια και κίνδυνοι και ε, πρέπει κανείς να τα αντιμετωπίσει αυτά τα πράγματα. Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι εάν πρέπει να ανοίξουμε ή όχι την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου που με απλά λόγια μιλεί για μη ευθύνη των πλατφορμών ηλεκτρονικής τεχνολογίας, για το περιεχόμενο δηλαδή που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Το αντιμετωπίζουμε αυτό με διάφορους τρόπους. Ζητούμε να αφαιρέσουν κηρύγματα μίσους, τρομοκρατικό περιεχόμενο, ε, παιδική πορνογραφία, αυτά, αυτά υπάρχουν νόμοι Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα που ίσως χρειάζονται βαθύτερη ανάλυση μπορούμε να εξετάσουμε κάποια α, θέματα οικειοθελούς δέσμευσης και να προχωρήσουμε και σε θέματα νομικής ευθύνης για το περιεχόμενο. νομοθέτημα δηλαδή για το ιδιωτικό, το ιδιωτικό τομέα που θα μπορούσε να προβλέπει ίσως κάποια ψηφιακή φορολογία. Δεν ξέρω όμως ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο που έχει στο μυαλό της η υποψήφια πρόεδρος και που θα το συζητήσει η επόμενη επιτροπή. Η παρούσα επιτροπή προχώρησε πολύ προσεκτικά σε ό,τι αφορά την ρύθμιση του ψηφιακού τομέα και εδώ μιλούμε βεβαίω πολύ για κράτο δικαίου, αλλά είναι και ο δημοκρατικό χώρο όπου μπορεί στο διαδίκτυο δηλαδή να εκφράσει την άποψή του καθένα. καθένας. Φανταστείτε τώρα να απαγορεύσουμε την ανωνυμία των ε, σχολιαζόντων. Θα ήταν σημαντικό πρόβλημα για του ανθρώπου αυτό. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να είμαι σύντομη, όμως ε, τέθηκαν πολλέ ερωτήσει και βέβαια η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο ψηφιακό ε, θέμα θα είναι ένα από τα σημεία κλειδιά και για την επόμενη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ρεαλιστικό να λειτουργήσει το 2020. Ναι, εφόσον εκλεγεί ο επικεφαλής σύντομα, διότι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, αλλά χρειαζόμαστε τον επικεφαλής. Ε, ετοιμάζουμε ε, την έδρα στο Λουξεμβούργο, την εξοπλίζουμε, έχουμε ρυθμίσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς. Μας επέκριναν οι χώρες ε, μέλη ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε και ότι αυτό δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά του ε, Συλλογικού Σώματος των Εισαγγελέων, College of Prosecutors. Θα δούμε. Βέβαια πρέπει και το Συμβούλιο να ρυθμίσει σε αυτά. Τώρα, data sharing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή η συζήτηση θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Πρώτα όμω, και ομιλώντα για την προστασία δεδομένων, αν αυτή καλύπτει τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, εδώ πρέπει να διευκρινιστούν πολλά πράγματα που έχουν σχέση με τι, μη μη ε, διότι υπάρχει μέσα στον κανονισμό GDPR διάκριση ανάμεσα σε εταιρείε οι οποίε έχουν το data processing, την επεξεργασία δεδομένων δηλαδή, ως βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουν, και εκείνες οι οποίες πολλούν, ξέρω ψωμί ή ε, εξοπλισμό κομμωτηρίων και που ε, δεν βγάζουν λεφτά από τη διαχείριση των ε, δεδομένων των προσώπων. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν πιο ευδιάκριτα για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις και γι' αυτό προωθεί την έγκριση των πιστοποιήσεων επίσης ε, κώδικες συμπεριφοράς για τις διάφορες ε, επιχειρήσεις κλπ. Για την μελέτη του Λονδίνου εδώ ομολογώ ότι δεν την έχω διαβάσει. Πρέπει να την εξετάσω. Η κυρία Σίπλ για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και τι, ποια είναι τα καθήκοντά μας εκεί. βέβαια είναι τεράστια αυτά. Όταν το 2014 ανέλαβα το χαρτοφυλάκιό μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αντιλήφθη ότι ο, το χαρτοφυλάκιό μου θα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικά ούτε φανταζόμουν ότι θα είναι τόσο αντιδημοφιλές, επίμαχο και επικίνδυνο, αλλά και ότι θα είναι αναγκαίο ε, να έχω, να υψώνω ε, ισχυρή φωνή για τα θέματα αυτά, για τα κηρύγματα μίσους στο διαδίκτυο, για τις επιθέσεις κατά διαφόρων προσώπων, όχι για αυτό που κάνουν, αλλά για αυτό που είναι διότι έχουν άλλο χρώμα ε, επιθερμίδας έχουν ε, διαφορετική γενετήσια, διαφορετικό γενετήσιο προσανατολισμό. Είναι αειδές αυτό που συμβαίνει πραγματικά, αυτά που συμβαίνουν σε ορισμένες ε, χώρες μέλη και online και offline. Και γι' αυτό πιέζουμε τις ε, ε, ηλεκτρονικές πλατφόρμες να αφαιρούν τα κηρύγματα μίσους, διότι αυτά οδηγούν και στην άσκηση βίας στην πραγματική ζωή. Βέβαια δεν μιλούμε μονάχα για την βία, και ξέρω ότι μιλήσατε ιδίω και για την διάκριση. Βλέπετε διάκριση, διακρίσεις να αυξάνουν σε διάφορους τομείς, όπως την εκπαίδευση. Και γι' αυτό θέλω να πιέσω για να γίνει, να εγκριθεί η οδηγία ίσων δικαιωμάτων τον Οκτώβριο στην ΕΠΣΚΟ. Χρειάζεται συζήτηση με τις χώρες μέλη και για το πιθανό κόστος, γιατί πάντοτε μιλούμε και για το χρηματικό και το επιχείρημα των χωρών μελών ήταν ότι το κόστος για τις διάφορες κατασκευές, για τις ε, ε, κυλιόμενες πολυθρόνες κλπ. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι μοναχά υπόθεση ενός είδους Υπουργείων. Και όταν ήρθαμε και στην εσωτερική συνεργασία, αν μα είπαν τότε χωρί μέλη, αυτό είναι σημαντικό, δεν μπορούμε απλώ να απόσχουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτά που είπατε βέβαια για την, τον αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφιλοφιλοφοβίας κλπ. Η οδηγία για την αστυνομία. Πρέπει να δούμε εάν υπάρχουν νέα στοιχεία και να σας απαντήσουμε γραπτός αν δεν έχετε αντίρρηση, ώστε να έχετε και μια πλήρη απάντηση και ενημερωμένη. Για θέματα ιδιωτικής σφαίρας, πώς θα διαπιστώσουμε αν οι επιχειρήσεις ακολουθούν τους κανόνες. Μα παρακολουθούνται και από το Υπουργείο Εμπορίου, τα Υπουργεία Εμπορίου, και δικαιοσύνης και την Federal Trade Commission που έχει ήδη απαγορεύσει την συμμετοχή ορισμένων επιχείρησεων στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας, το σύστημα λειτουργεί πιο ενεργά από ό,τι στις αρχές του. για το άρθρο 7, πιο ξεκάθαροι κανόνες και τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό. Όταν μιλεί η Επιτροπή για την πολωνική υπόθεση, όπου το άρθρο 7 έγινε επίκλησή του δηλαδή για πρώτη φορά, τα κρατήσαμε εμείς στην Επιτροπή για πολύ καιρό ε, στους κόλπους της Επιτροπής. Κάποια στιγμή όμως, μετά από επιστολές και επιστολές, ε, έγινε προφανές ότι πρέπει να καταλήξει στα τραπέζια των Υπουργών. Και έφτασε τελικώς στα γραφεία του Συμβουλίου. Συζητήσεις χρήσιμες και σημαντικές. Με ρωτούν καμιά φορά οι δημοσιογράφοι Μα πώς, λειτουργεί το άρθρο 7 αφού δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Και όμως και η συζήτηση είναι σημαντική. Και την προηγούμενη εβδομάδα στο Ελσίνκι, η παρουσία και του κ. Αγγιλάρ, έγινε η συζήτηση αυτή. Οι Υπουργοί Δικαιοσύνη πρέπει επίση να αρχίσουν να συζητούν το θέμα αυτό, γιατί πρόκειται για κράτο δικαίου σε χώρα μέλο και είναι ο τομέα τη δικαιοσύνη. Και τελικώ αυτοί πληρώνουν το τίμημα, διότι αν υπάρχουν κενά στο κράτο δικαίου σε κάποιε χώρε μέλη, τότε πάβει να λειτουργεί το σύστημα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Συλλήψεων, η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αναγνώριση των αποφάσεων, αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων δικαστηρίων. Πρόκειται δηλαδή για σημαντικό, σοβαρό, συστημικό πρόβλημα που πλήττει ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό και το συζητήσαμε και θέλουμε να καταλήξουμε σε κάποιε αποφάσει πιο πρακτικής μορφής και θυμηθείτε ότι το Συμβούλιο Δικαιοσύνη, Υπουργών Δικαιοσύνης, ε, μακρηγόρο κάπως, ναι, είναι το ερώτημα, είναι πολιτικό το θέμα ή είναι καθαρά νομικό. Εγώ νομίζω ότι έχει και τις δύο αυτές πλευρές. Και γι' αυτό και τα δύο ε, Συμβούλια ε, Δικαιοσύνης και Γενικών Υποθέσεων πρέπει να εγκύψουν. Η ε, κυρία Σοφίντ Φέλτ για την ε, για τα θέματα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Από τα πιο σημαντικά μας προβλήματα. Η Ευρωπόλ μόλις πρόσφατα εκτιμά ότι κάθε χρόνο το ξεπλημένο βρώμικο χρήμα φτάνει στο ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, δηλαδή 1% ολόκληρου του ε, ε, ε, εθνικού προϊόντος των χωρών μελών, 150 δις. Και όλα είναι και θέματα βέβαια διαφθοράς, ε, διαμεθοριακά διαδίκτυα οργανωμένων εγκληματιών. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε. Πάλι αν μια, δυο, τρεις χώρες αμελούν τα καθήκοντά τους θα καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα στην Ευρώπη και ήδη βρίσκεται σε κίνδυνο γιατί βλέπουμε τέτοιες ε, υποθέσεις να αναφύονται και γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή επιτήρηση, μιλούμε για ανάγκη να υπάρχει κανονισμός, διότι μέχρι τώρα ισχύουν οδηγίες στο χώρο μόνο του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο. Και υπάρχουν τόσο διαφορετικέ προσεγγίσεις από τι χώρε μέλη και με ε, εντελώ αναξιόπιστα αποτελέσματα. ενώ χρειάζεται ευρωπαϊκό όργανο για την επιτήρηση. Αυτά όμω θα τα αποφασίσει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Δηλαδή το νέο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, η αναγνώριση του κράτου δικαίου, ναι, δεν είναι επαρκή. Ανέμενα την κριτική αυτή, το, συζητούμε σε βάθο. Υπάρχουν κεφάλαια όπου η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ε, και η εισαγγελία είναι ένας πυλώνας μόνο. Υπάρχει και ο χώρος της κοινωνίας των πολιτών. Η ελευθερία λόγου και η ελευθερία τύπου. Οι κρατικέ διοικήσεις που δεν λειτουργούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Ε, είναι πολύ ευρύτερο λοιπόν το θέμα. Και δεν μπορούμε σε μια ανακοίνωση να τα περιλάβουμε όλα. Θέλαμε να επισημάνουμε τον μηχανισμό που θέλει και το Κοινοβούλιο και γιατί δεν βάζουμε τώρα και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, διότι οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι εάν η ετήσια αξιολόγηση φέρει τέτοια αποτελέσματα που να έχουν νομικές επιπτώσεις, να αρχίσουν δηλαδή προσφυγές για παραβιάσεις κλπ. Θα πρέπει να έχουμε την πιο ισχυρή δυνατή νομιμοποίηση της αξιολόγηση αυτή. Άκουσα και μετά την ερώτηση αυτή από κάποιον. Πώς θα μετρήσουμε δηλαδή την ισχύ του κράτους δικαίου στις χώρε μέλη. Μα με αυτό το ζήτημα συνδέεται. Έχουμε 28 διαφορετικά συνταγματικά συστήματα. Έχω ξεπεράσει κατά 15 λεπτά, όχι 5 λεπτά έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Όμως υπάρχουν και τόσο πολλοί άλλοι που θέλουν να παρέμβουν που θα είμαστε ευγνώμονες αν μπορέσετε να εξοικονομήσετε όσο το περισσότερο χρόνο για να ακούσετε και τα άλλα μέλη. Θα μου πούν και άλλες ερωτήσεις για ε, το κράτος δικαίου, άρα μπορώ να τα πω και μετά αυτά που θέλω να πω. Ε, το Ταμείο για την Επίρρηση Διαφορών θα το εξετάσω πάλι και μπορούμε να σας απαντήσουμε διμερώς αν θέλετε. Πρέπει να μιλήσω με τις υπηρεσίες μου πρώτα. Νομίζω πάντως ότι κάναμε ό,τι μπορούμε για το νέο πρόγραμμα ε, αξιών και δικαιωμάτων και το συζητούμε πάντως αν θέλετε. Άλλο τίποτε. Η κυρία Ράιντκε τόσα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Θα επανέλθω. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Λοιπόν, 21 ακόμη θέλετε το λόγο. 1,5 λεπτό έκαστος λοιπόν, για να έχουμε και χρόνο μετά, ώστε η ε, Επίτροπος να απαντήσει σε αυτό το δεύτερο γύρο. Είναι προφανές ότι θα ξεπεράσουμε το προγραμματισμένο μας χρόνο και θα χρειαστεί να αναβάλουμε κάποια θέματα όπως το 8 που είναι η, εξέταση του πίνακα επιδόσεων για τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, 1,5 λεπτό ο καθένας ώστε να μπορέσετε όλοι να πάρετε το λόγο. Κύριο Σασαλέχος. Presidente, muchas ευχαριστώ πολύ. Θέλω να μιλήσω για την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων. Φαίνεται πως υπάρχει ε, πρόβλημα. Αυτό σημαίνει πως η εφαρμογή του ευρωεντάλματος δεν έχει εδρεωθεί για, παρότι είναι η πιο έντονη έκφραση της ε, δικαστικής δικαιοσύνης, δεν θέλω τώρα να θέσω σε προφυσβήτηση τα όσα λέει το άρθρο 2, αλλά θα ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις για να καταλάβω πώς το σκέφτεσαι. Οι πιθανές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να μπουν στην διαδικασία του εντάλματος, ώστε από τη μια πλευρά να εγγυηθούμε την κατάλληλη αντιμετώπιση των ε, ενταλμάτων ε, από όλα τα δικαστηρία. Ας πούμε υπάρχει ένα πρόβλημα ενός, ε, του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά ενός κράτους μέλους ε, και έπειτα να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης αποφεύγοντας την εξοδαφικότητα τον, ε, μάλλον την εξαίρεση των δικαστηρίων που λαμβάνουν ε, τις εντολές αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Καθώς μίλησε ο κύριος Σανθελέχος, κάποιοι άλλοι σηκώσατε τις ε, κάρτες σας. Οπότε θα πρέπει μάλλον να κλείσω τον κατάλογο μιλητών τώρα. για τους νεοεκλεγέντες θα πρέπει να ξέρετε ότι η Επίτροπος είναι πάντοτε πρόθυμη να δώσει και γραπτές απαντήσεις για όσους δεν ε, ικανοποιήθηκαν πλήρως από τις απαντήσεις που έλαβαν. Θα υπάρξει λοιπόν και γραπτή απάντηση. Turn for Mr. Bitanov. Ο κύριος Μπίτανοφ τώρα. Sorry. As a newcomer. Ε, συγγνώμη, είμαι και νέος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα από την ανακοίνωση της προηγούμενης εβδομάδας, θα υπάρχουν ετήσιες εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος και αυτό θα αντικαταστήσει τον μηχανισμό που υπήρχε μόνο για Βουλγαρία και Ρουμανία. Καλωσορίζω αυτήν την απόφαση γιατί έτσι θα καταργηθούν αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ε, είχαν ειδική αντιμετώπιση για πάρα πολύ καιρό και βεβαίω είναι εμφυλεγόμενα τα αποτελέσματα, τουλάχιστον στη Βουλγαρία. Οι Βουλγαροί πολίτες ε, δεν εμπιστεύονται ιδιαίτερο στην δικαιοσύνη. Η Βουλγαρία ε, έχει ε, μία από τι τελευταίε θέσει στην κατάταξη. Ο μηχανισμός αυτός ε, κράτους δικαίου ε, δεν είναι πάρα πολύ αποτελεσματικής και κάποια κράτη-μέλη το χρησιμοποιούν αυτό ως δικαιολογία για να μην επιτρέψουν στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να μπουν στη Σέγγεν. Παρά το ότι είχαμε κάποιες θετικές εκθέσεις ε, στο παρελθόν, το ερώτημά μου είναι πότε θα καταργηθεί το παλαιό σύστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιούρεβα. Επίτροπε Γιούροβα. Ε, ε, πάντοτε είναι ευχάριστο να σας ακούμε και σας ευχαριστώ για την εργασία που έχετε κάνει με όλα αυτά τα χρόνια. Μιλήσαμε για αμοιβαία εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα μέσα που δημιουργούν αυτή την εμπιστοσύνη και την δικαστική συνεργασία στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος ε, Θανθαλέχος. Πράγματι, το 2014 ήδη το Ευρωκοινοβούλιο είχε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι ορισμένα από τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών έβγαζαν ε, ε, εξέδιδαν ε, ευρωπαϊκά εντάλματα για διάφορα ίσονα σημασία αδικήματα, όπως α πούμε, ε, μάλλον, αλλά ότι τελικά δεν εφαρμόζονταν. Έχουμε μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό ένταλμα από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ωστόσο, το δικαστήριο ενός κράτους μέλους, ε, ενός κράτους μέλους ε, μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση του εντάλματος λόγω προβλημάτων που υποτίθεται ότι βρίσκει. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ευρωπαϊκά κριτήρια. Να μην μπορούν τα κράτη-μέλη να αποφύγουν να εφαρμόσουν αυτά τα ε, ευρωπαϊκά κριτήρια του εντάλματος, του ευρωπαϊκού εντάλματος. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν, αυτούς τους τελευταίους μήνες εσείς θα πρέπει να ευαισθητοποιήσετε ευαισθητοποιήσετε τον διάδοχό σας ή την διάδοχό σας ώστε να βελτιωθεί η εφαρμογή του ευρωεντάλματος γιατί ε, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την ευρωπαϊκή συνεργασία στα, θέματα ελευθεριών, θεμελιδων δικαιωμάτων γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η αρχή της ισότητας. Χρειάζεται λοιπόν να ενισχυθεί και να μεταρρυθμιστεί αν είναι δυνατόν αυτό αυτό και άλλα μέσα συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να αφήσετε κάτι ήδη έτοιμο στο διάδοχό σας. Ευχαριστώ. Μοράλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επιτροπέ, επιτρέψατε μου να σας ευχαριστήσω για την συνεργασία που είχαμε στην προηγούμενη θητεία. Γνωρίζουμε ότι προσπαθείτε να αποφύγετε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά πέρα από την δίτη ποιότητα προϊόντων, τροφίμων ε, κτλ. Υπάρχει και ο μηχανισμός CVM που είναι αρμοδιότητός σας. Πρόκειται εξορισμού για δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ισχύει μόνο για δύο κράτη-μέλη. Εδώ και πολλά χρόνια η Βουλγαρία και η Ρουμανία ακούνε υποσχέσεις ότι ο διακριτικός αυτός ε, μηχανισμός θα καταργηθεί. Ε, είχαμε κάποιες θετικές εκθέσεις της Κομισιόν, ε, μεταρρύθμιση, πολιτική βούληση των κρατών μελών κτλ. Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε υποσχεθεί πολλά και ότι θα καταργηθεί η παρακολούθηση αυτή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η θητεία της Κομισιόν. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί παρά το ότι η Βουλγαρία πληρεί τα κριτήρια. Επιπλέον, ένας νέος μηχανισμός παρακολούθησης του κράτους δικαίου έχει αναφερθεί για πολλές περιπτώσεις που θα ισχύσει για όλα τα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πλέον η ανάγκη αυτού του μηχανισμού. Ε, η ερώτησή μου είναι η εξή. Η Κομισιόν παρουσίασε την ερώτησή τη για το θέμα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Η von Φοντερ Λάιεν υποσχέθηκε προσωπικά ότι θα εισαχθεί ένας τέτοιος ε, μηχανισμό. Πότε λοιπόν θα καταληφθεί ο μηχανισμό αυτό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία μπορούμε να αναμένουμε ότι η έκθεση του Σεπτεμβρίου θα είναι η τελευταία. Κύριε Ιζερέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Ω ε, μέλο τη ομάδα κατά του ρατσισμού θα ήθελα να αναφερθώ στα εγκλήματα μίσου. Ε, αναφερθήκατε λίγο, αλλά θα ήθελα να πάω λίγο πιο πολύ σε βάθο Παρά τι προσπάθειε των κρατών μελών, τα στοιχεία δείχνουν ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Κάποια βήματα βεβαίως έχουν ληφθεί, όμως ε, δεν αρκούν και είμαι πεπισμένη ότι απαιτείται νέα νομοθεσία έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα εγκλήματα μίσους. Έχουν αναφερθεί συγκεκριμένες ελλείψεις από τις αρμόδιες ΜΚΟ και την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης. Είναι η έλλειψη προστασίας ε, των θυμάτων, ε, ε, θυμάτων που πέφτουν ε, θύματα των σεξουαλικής ταυτότητας. Το ερώτημά μου θα μπορούσε να επεκταθεί λοιπόν ο ορισμός ρατσισμού και ξενοφοβίας για να περιλαμβάνει την ταυτότητα φίλου και τα λοιπά και μπορείτε να μας ενημερώσετε εάν υπάρχουν ε, κάποιες ε, διαδικασίες σε παραβάσεις κατά κρατών μελών που δεν έχουν ε, εφαρμόσει τις αποφάσεις σωστά και δεύτερον κατά το οποίο αφορά την πιο οριζόντια οδηγία που είναι μπλοκαρισμένη αυτή τη στιγμή όπως είπατε στο Συμβούλιο μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το πώ έχει αυτή η νομοθεσία. Αν δεν αλλάξει τίποτα στο Συμβούλιο μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα υποβάλλετε νέα πρόταση και θα ζητήσετε από το Συμβούλιο να την εγκρίνει. Σύμφωνα με την τακτική νομοθετική διαδικασία έτσι ώστε να εμπλακεί και το Κοινοβούλιο σε νομοθέτηση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ε, παρακαλώ προσπαθήστε να περιοριστείτε στο 1,5 λεπτό για να μιλήσουν όλοι. Κυρία Κέλλερ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ ε, για το χρόνο σας ε, ε, που είστε διαθέσιμοι και που μας αναφέρατε, να μας δώσατε αναφορά για τις δράσεις σας. Δύο ερωτήσεις. Όσον αφορά τα μέτρα κατά του ξεπλήματος χρήματος, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιες, πώς συνεργάζεστε με τον ΩΣΑ και άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, διότι το ξέπλήμα χρήματος είναι ένα θέμα παγκοσμιοποιημένο. Δεύτερη ερώτηση, προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να μας εξηγήσετε στο τέλος ε, μια, μιας θητείας όπου, είστε, όπου ήσασταν ιδιαίτερα διαδραστήρια για αυτό το θέμα. Στο μέλλον, τι θα πρέπει να κάνουμε για να με βελτιώσουμε την ε, προστασία δεδομένων και να βελτιώσουμε και την ε, ζωή των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρέγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αφορά την νομοθεσία περιψιακών υπηρεσιών. Είχαμε κάποιε πληροφορίε στα ΜΜΕ για το τι θα μπορούσε να περιέχει σύμφωνα με τα σχέδια τη Γενική Διεύθυνση Connect και ανησυχώ ιδιαίτερω για το ότι η νομοθεσία αυτή θα μπορούσε να κάνει τις πλατφόρμες αυτές ένα είδος αστυνομία ή λογοκοριτών του διαδικτύου. ή να δημιουργήσει τα διάφορα φίλτρα που γνωρίζουμε ότι κάνουν πολλά λάθη και βεβαίω ε, τα πολύ στενά χρονικά πλαίσια για την αφαίρεση του περιεχομένου θα μπορούσαν να τιμωρήσουν τις μικρές ε, επιχειρήσεις. Μπορείτε λοιπόν να μας διαβεβαιώσετε ξανά για το ποια είναι η θέση σας ε, ειδικά στον αφορά τα φίλτρα. Δεύτερη ερώτηση. Στο πλαίσιο των σχετικό, της σχετικής αυτής νομοθεσίας ε, θα μπορούσατε να δεσμευτείτε για ένα δικαίωμα ανώνυμης χρήσης ε, του διαδικτύου για να μην υπάρχει κίνδυνος κλοπής ταυτότητας. Ε, ήδη υπάρχει αυτό το δικαίωμα στη Γερμανία όπου είναι τεχνικά δυνατό. Μπορούμε να το έχουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τρίτη μου ερώτηση αφορά την διασυνδεσιμότητα. Ένα στοιχείο της σχετικής νομοθεσίας θα μπορούσε να είναι η διασύνδεση των υπηρεσιών ε, μήνυμάτων και κοινωνικών δικτύων έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αλλάζουν και να έχουν δικαίωμα επιλογής. και να πάνε σε μια πλατφόρμα που θα προστατεύει καλύτερα τα δεδομένα τους. Θα ήσασταν υπέρ. Ευχαριστώ κυρία Σόφση. Ο κύριος Σόφση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω την Τσεχική τη γλώσσα μου. Πρώτα απ' όλα, σας υπενθυμίζω ότι ήσταν εδώ πέρα ε, πριν από λίγου ε, μήνε ε, για να μιλήσετε για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Μιλάμε για διαρροή δεδομένων εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών και είπατε ότι θα δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι έχει γίνει, πώς πάει η έρευνα και εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να αναμένουν ότι θα επιβληθεί πρόστιμο στο Facebook. Δεύτερη ερώτηση. Κάπως παρόμοια, αλλά εξίσου σημαντική είδαμε μόλις το σχέδιο προϋπολογισμού. Ποια είναι η άποψή σας ε, για το ότι η Κομισιόν αφενός ε, δεν λέει ότι θα πολεμήσει την τρομοκρατία, την ε, διακίνηση ανθρώπων και απ' την άλλη υπάρχουν περικοπές σε 52 θέσεων προσωπικού σε Europol και Eurojust. Τόσο μεγάλες περικοπές ώστε το αργότερο τον Οκτέβριο, πλέον δεν θα είναι επιχειρησιακέ και δεν θα μπορούν να συνεργαστούν σε περιπτώσει οργανωμένου εγκλήματος. Σας ευχαριστώ. Κινίτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τον νόμο για την καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος. Εγώ θα ήθελα, εάν θα μπορώ, να γνωρίζω αν μπορείτε να μας εγγυηθείτε τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και της ε, Κεντρικής Τράπεζας που έχει ένα γενικότερο υποπτικό ρόλο. Μετά, για να αλλάξω εντελώ θέμα, μία άλλη ερώτηση. Αναφέρομαι στην σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης, η οποία μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ στην ε, θητεία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποια μέτρα θα μπορούσε να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τα κράτη-μέλη στην συγκεκριμένη εφαρμογή τη συνθήκη. Γιατί γνωρίζουμε ότι πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν κάνουν τίποτα ε, ούτε αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το θέμα και ποια μέσα του ευρωπαϊκού δικαίου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία των θυμάτων ε, βίας ε, έμφυλης και επίσης και των ε, παιδιών ε, που επίσης ε, μπορούν να αποκτήσουν τραύματα που θα τα σημαδέψουν για όλη τη ζωή. Επίσης, αν θα μπορούσατε να σκεφτείτε κάποιες άλλαγες στην Οδηγία 29 του 2012 για το σύστημα προστασίας των θυμάτων για να ενισχύσουμε την προστασία, όπως σας είπα, των ανηλίκων, των παιδιών στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Φράντς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ εκ καρδίας ε, κυρία Γιουροβά για τη δουλειά που έχετε κάνει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς και πότε σκοπεύει η Κομισιόν να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχετικού πλαισίου του στρατηγικού σχεδίου για την διακριτική μεταχείριση των Ρωμά και την καταπολέμηση του αντιτσιγκανισμού επιτέλους πρέπει να υπάρξει ένας δεσμευτικός χαρακτήρας, γιατί όπως γνωρίζετε υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη οι οποίοι υφίστανται διάκριση, όπως ο Γκάνι Ράμα, ένας Ρώμ στο Κοσφοπέδιο ο οποίος εδάρει στην Πριστίνα. Ένας άλλος ο οποίος πυροβολήθηκε στο σπίτι του στη Βουλγαρία, στην ε, Ιταλία τους βάζουν φωτιά στα σπίτια τους, όπως και στο Ούλμ στη Γερμανία υπήρξε μια εμπριστική επίθεση. Η Ρωμά είναι η ομάδα εκείνη η οποία υφίσταται τις χειρότερες επιθέσεις, βίαιες επιθέσεις ε, και έχουν ε, τραγικές συνθήκες στέγασης ε, και εκπαίδευση κτλ. Δεν υπάρχει πρόβλημα Ρωμά, υπάρχει πρόβλημα ρατσισμού και πρέπει να το σταματήσουμε επιτέλους. Σας ευχαριστώ κύριε Φέστ. Ναι, καλημέρα σας κυρία Γιούροβα. Δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν απαντάτε σε ερωτήσεις μόνο των αριστερών, αλλά τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου η εντύπωση. Δεν απαντήσατε στους κυρίους Σταρντίνο και Ποκατσίνη αυτή η μεταχείριση των ερωτήσεων πώς συμβιβάζεται με το ότι θα πρέπει να είστε υπερκομματικοί ως Επιτροπός. Δεύτερον, μια που είμαι μέλος στην Επιτροπή των Γυναικών, γνωρίζετε το ότι σε μέλη στα οποία έχουν υπογράψει την σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης αν έχει υπάρξει μια στατιστικά καταγεγραμμένη μείωση της ε, οικογενειακής βίας ή ε, εξακολουθεί να έχει το ίδιο ύψος ε, και, όπως και πριν, την ίδια έκταση όπως και πριν. Σας ευχαριστώ κύριε Μπουρέκα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, πρώτα κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την καλή δουλειά που κάνατε τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχουν φιλόδοξες και αναγκαίες πολιτικές, πρέπει να συνεχιστούν. Τώρα, πρώτο, βία κατά γυναικών και οικιακή βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και να μπορέσει να ε, συνυπογράψει την ε, διάσκεψη, την, ε, μάλλον την σύμβαση της Ισταμπούλ της Κωνσταντινούπολης και το άρθρο 83 της συνθήκης να αναθεωρηθεί. Η υποψήφια πρόεδρος της Κομισιόν στηρίζει την προσέγγιση αυτή. Ε, είναι διατεθειμένη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να εργάζεται ήδη. Δεύτερο, οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων. Δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για τις ανισότητες σε βάρος ε, αναπήρων και ε, προσώπων LGBTI. Προσπαθήσατε να αναθεωρήσετε την οδηγία το 2014 και σας ευχαριστούμε πολύ που το πράξατε αυτό. Τώρα όμως είμαστε 2019 και έχει έρθει η ώρα πια να το κάνουμε. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορούμε να κάνουμε πριν ήδη να αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μαγκίτ, ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειάζεται ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Αναγκαίο αυτό για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού συστήματο. Όμω, δεν εφαρμόζονται οι κανόνε με τον ίδιο τρόπο σε όλε τι τράπεζε και σε όλες τις χώρες μέλη. Δεν μπορούμε ε, να αφήσουμε να υπάρχουν αδύναμα σημεία στο ευρωπαϊκό σύστημα που να τα εκμεταλλεύονται οι εγκληματίε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ενθαρρύνουμε όλε τι χώρε μέλη να εφαρμόσουν του κανόνε αυτού στι επικράτειέ του. Και τι θα πείτε στην διάδοχό σας και στη νέα πρόεδρο τη Επιτροπή για να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό. Και τέλο, για εγκλήματα μίσου. Υπάρχει σχετική νομοθεσία, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Όμω, μόνο ένα μικρό κλάσμα των ε, θυμάτων καταγγέλει τέτοια εγκλήματα. Και πολύ συχνά η αστυνομία δεν τα αντιλαμβάνεται καν αυτά ως, ως εγκλήματα μίσους. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε και να ε, επιμείνουμε ώστε όλες οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρώπης να έχουν τον πλήρη εξοπλισμό, δηλαδή ε, όχι μόνο τεχνικό αλλά και ηθικό διοντολογικό, για να αντιμετωπίζουν τα πράγματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ βρίσκομαι. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας. Είμαι νέο μέλος <clears throat> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκφράζω την ελπίδα και στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα συνεχίζω στα αγγλικά. Δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στις ίσες ευκαιρίες και στην ε, δικαιοσύνη. Και στην δική μου εκλογική εκστρατεία, για να εκλεγώ δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήταν και μπήκε και το θέμα των ε, διπλών προδιαγραφών ε, εμπορευμάτων που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά. Θέμα το οποίο είχε θέσει και ο κ. Ιούνκερ προδιετία. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό και σα ρωτώ ποια είναι η αξιολόγηση που κάνετε των επιτευμάτων της προσπάθειας αυτής για να εξασφαλίσετε μια ε, δικαιοσύνη στην ενιαία αγορά και να έχουν όλοι οι καταναλωτές σε όλες τις χώρες μέλη ε, πρόσβαση στα ίδια αγαθά ε, ίδιας ποιότητας δηλαδή. Και τώρα για τον κανονισμό GDPR. Ποιες είναι οι επιπτώσεις ενδεχομένως ε, για τον GDPR εφόσον ε, γίνει ε, άτακτο Brexit. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάρλεϊ. Καλώς ήρθατε κυρία Γιούροβα. Θα ήθελα να επανέλθετε στο κράτος δικαίου και να τονίσετε περισσότερο αυτά που θέλετε να πείτε. Ήδη σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε, ότι δηλαδή δεν είναι μονάχα δικανικό θέμα, είναι και ζήτημα πολιτικό. Το ακούσαμε αυτό και από την κυρία Φοντελάιν. Είναι και ζήτημα μηδέας εμπιστοσύνη. Και ποιε θα είναι οι επιπτώσεις αυτής. Μπορείτε να μιλήσετε λίγο για τις επιπτώσεις. Και ιδίω για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Ευχαριστώ. Λαγοδίνσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Μιλούμε για το κράτος δικαίου. Όμως, επισημαίνω ένα θέμα. Μιλούμε αφενός για το κράτος δικαίου, αφετέρου μιλούμε για ηλεκτρονικές αποδείξεις και ζητήματα ψηφιακά. Αυτά όμως πρέπει να είναι όλα μαζί, να μπουν όλα μαζί, γιατί αν εξετάζουμε την κατάσταση των ηλεκτρονικών αποδείξεων, τώρα, υπάρχουν ε, κατάφορες παραβιάσεις του κράτους δικαίου εκεί. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ο κανόνας, της, διαδικαστικός κανόνας δηλαδή ηλεκτρονικών αποδείξεων, όπως το έχετε προτείνει εσείς, σημαίνει ότι αυτομάτως δίνουμε ηλεκτρονικές αποδείξεις κατ' έτοιμα άλλων χωρών. Ταυτόχρονα, στην περίπτωση του εντάλματος συλλήψεως, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν συμμορφώνονται στις επιταγές του κράτους δικαίου. Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό. Δεν τα βλέπουμε αυτά ε, στην οδηγία e-evidence. Και υπάρχει και θέμα ταξινόμησης προσωπικών ε, δεδομένων. Που η νέα ρύθμιση είναι τελείως διαφορετική από οτιδήποτε στο παρελθόν και προκαλεί σύγχυση. Το ίδιο για την συνθήκη μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Τι θα κάνετε εκεί, για παράδειγμα, με παραβιάσεις του κανονισμού GDPR και ιδίω των άρθρων 6 και 48. Εν τέλει δηλαδή, rule of law και ψηφιακά. Και να απαντήσω στον ακροδεξιό που μίλησε πριν, υπάρχουν σαφή πρότυπα του κράτους δικαίου. Δεν μιλούμε για κράτος δικαίου σαν κάποια όριστη έννοια. Δεν ενδιαφέρεται καν να με ακούσει από ό,τι βλέπω. Διαβάστε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μιλούμε για ξεκάθαρες αρχές κράτους δικαίου. Και μην παριστάνετε ότι δίθεν το κράτος δικαίου είναι μια αφηρημένη έννοια. Ευχαριστώ. Τρουγκάροφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κυρία Επιτρόπε. Σας ευχαριστώ πρώτα για τη σκληρή δουλειά που έχετε κάνει σε όλη την θητεία σας. Και ιδιαίτερος σας ευχαριστώ με την ευκαιρία για την προσπάθεια που κάνατε για την χώρα μου, τη Ρουμανία. Και είμαι βεβαία ότι πολλοί Ρουμάνοι και πολλές Ρουμάνες εκτιμούν το έργο σας. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι ελπίζω ότι ο νέος μηχανισμός κράτους δικαίου θα είναι τουλάχιστον το ίδιο ισχυρό όπως ο προηγούμενος για όλες τις χώρες μέλη με σαφή κριτήρια. Και για τη Ρουμανία ο CVM μας κράτησε μακριά από το Σέγγεν αλλά η πολιτική αστάθεια και οι πρόσφατες επιθέσεις κατά του κράτους δικαίου από την ίδια τη ρουμανική κυβέρνηση τα επιδίνωσαν τα πράγματα. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτο, πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχει κάποια πρόοδος. Διότι η απόφαση λήφθηκε το 2014. Πού βρισκόμαστε τώρα. Δεύτερο, πλαίσιο του κανονισμού GDPR. Χθε η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της νέας αυτής νομοθεσίας τα περασμένα χρόνια. Στην Ρουμανία έχουμε μια κατάσταση όπου με την κατάχρηση της νομοθεσίας αυτής φημώνουν τον τύπο. Και εκεί διαμορφώνονται δύο καταστάσεις. Αφενός, ο GDPR εφαρμόζεται από εθνικές αρχές για να αναγκάσουν Ερευνητέ δημοσιογράφου να αποκαλύψουν τι πηγέ του, πολύ σοβαρή κατάσταση. Και δεύτερο, δεν του χορηγούν δημόσιου χαρακτήρα πληροφορίε, πάλι επικαλούμενε οι αρχέ, δηλαδή, το GDPR. Ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε Πίτροπε, σε ερώτηση που σας είχαμε κάνει πρόσφατα για το πώς τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απαράδεκτη αντικομουνιστική δίωξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Πολωνία, τη εφημερίδα του και τη συντακτική του Επιτροπής, Επιχειρήσατε να απαντήσετε ισχυριζόμενοι ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι στα κράτη-μέλη έχουν, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει νομοθεσία για την απαγόρευση χρήση συμβόλων του κομμουνιστικού παρελθόντο και ότι η Επιτροπή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τη ήταν πάντα σταθερά προσιλωμένη στη μνήμη σχετικά με ολοκληρωτικά καθεστώτα, λέτε. Ε, κάθε κράτο μέλο έχει βρει τη δική του προσέγγιση για να θυμάται την ιστορία του. Κυρία Γιούροβα, η εξίσωση του κομμουνισμού με το τέρα του φασισμού είναι και ανιστόρητη και ανυπόστατη. Τα περί ολοκληρωτισμού δεν έχουν βάση γιατί πάνω απ' όλα ο φασισμό και η αστική δημοκρατία έχουν κοινή οικονομική βάση την καπιταλιστική ιδιοκτησία. Και όχι βέβαια ο σοσιαλισμό που η εξουσία είναι στα χέρια του λαού. Την ίδια ώρα, μάλιστα, που η Ευρωπαϊκή Ένωση σηκώνει θόρυβο στην Πολωνία για την κατάσταση στον τομέα τη δικαιοσύνη, γεγονό που εκφράζει συντηνόμενε αντιθέσει μεγάλων συμφερόντων εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πλήρη κάλυψη στου αντικομουνιστικού νόμου και τι αντικομουνιστικέ διώξει στην ίδια χώρα. Τι έχετε επίση να πείτε για το ότι στι 16 Ιούλη το Συνταγματικό Δικαστήριο τη Ουκρανία επέβαλε την απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματο Ουκρανία. Τα περιμία αρμοδιοτήτων σα στα κράτη-μέλη σε άλλε χώρε είναι υποκριτικά, γιατί στηρίζετε και χρηματοδοτείτε εκστρατείε με, αντικομ... αντικομουνιστικό και ανιστόρητο περιεχόμενο, όπω το πρόγραμμα Ευρώπη για του πολίτε σε κράτη-μέλη, ενώ αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι πολιτικέ ελευθερίε μόνο ω όργανο για επεμβάσει και εξασφάλιση συμφερόντων όπου υπηρετεί και παρεμβαίνει στι εσωτερικέ υποθέσει κρατών σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Επικροτεί τον αντικομουνισμό ω συνέχεια τη αντιλαϊκή αντεργατική πολιτική. Απέναντι σε αυτά λοιπόν σα λέμε ο αντικομουνισμό θα πέσει στο κενό, κάτω τα χέρια από του κομμουνιστέ, του Πολωνού, του Ουκρανού, τι χώρε τη Βαλτική και απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσουν όλε οι αντικομουνιστικέ διώξει. Ευχαριστώ. Κυρία Γιόντσεβα, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά την ε, Βουλγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε ότι υπάρχει ε, διαφορά υψηλού επίπεδου και ενώ η Κομισιόν τα σημειώνει αυτά, η ε, διαφθορά γιγαντώνεται. και δεν ε, ελέγχεται, δεν ελέγχονται καθόλου ε, οι εισαγγελείς στη Βουλγαρία οι οποίοι δρούν με βάση πολιτικές εντολές. Έχετε συστάσεις ε, για τις εισαγγελίε και λέτε ότι δεν θα πρέπει να υφίστανται κανέναν έλεγχο. Κάτι άλλο. Προσφάτως στη Βουλγαρία είχαμε ένα χακάρισμα των δεδομένων της εφορίας τα δεδομένα εκατομμυρίων φορολογούμενων πολιτών διέρευσαν. Και κάποια ΜΜΕ είπαν ότι ε, ολόκληρη χώρα πλέον, τα δεδομένα ολόκληρη χώρας διέρευσαν. Ποιος θεωρείτε ότι είναι υπεύθυνο για τα κενά στην ε, πολιτική ασφαλείας των πληροφοριών της χώρας και θα επηρεάσει αυτό την ένταξή μας Σέγγεν. Σας ευχαριστώ για την ε, τεχνητή νοημοσύνη έχετε αρχίσει να κοιτάτε αυτό το ζήτημα που πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι θα επηρεάσει ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τους καταναλωτές. Μάλιστα, έτσι. Σύντομα και απλά. Οπότε τελευταίος ο κύριος Γιάκη. Έγινε πολλής λόγος για το κράτος δικαίου και τις αρχές ε, του, αλλά χωρίς να μπούμε στη λεπτομέρειε, όλα ήταν πολύ επαγγελματικά, αλλά ε, κυρίως με πολιτικές αποχρώσεις. Κάθε φορά που ρωτώ τι σημαίνει η παρατβίαση του κράτους δικαίου, μου λένε ότι ο διορισμός των δικαστών στην Πολωνία είναι πολιτικοποιημένος. Πώς λοιπόν γίνεται αυτό. Έχουμε ένα συμβούλιο που αποτελείται από δικαστές και που ορίζει τον, τον νέο δικαστή πώς ορίζονται οι δικαστές στη Γερμανία. Υπάρχουν πέντε δικαστήρια για τα οποία μια επιτροπή στην οποία συμμετέχουν με πολιτικοί και υπουργοί που εκλέγει τους δικαστές. Στην Πολωνία οι δικαστές ορίζονται από τους ε, συναδέλφους τους, ενώ στη Γερμανία οι πολιτικοί ορίζουν τους δικαστές και εκεί δεν θεωρείται πως είναι αυτό πολιτικοποιημένο. Κύριε Επίτροπε, μπορείτε να μπείτε σε λεπτομέρειες και να απαντήσετε σε αυτό το επιχείρημα που σας υποβάλλω, γιατί εδώ γίνεται πολλής λόγος και για γενικότητες, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουμε ε, ε, ε, ε επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ είμαι νοεκλεγίσα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Γιούροβα που μας ε, μίλησε για τα ε, δικαιώματα των γυναικών. Η ερώτησή μου είναι σύντομη και σαφής. Φαντάζομαι πως δεν είναι εύκολο έργο να συνεργάζεται κανείς με όλα τα κράτη-μέλη σε σχέση με την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών. Αυτό που θα ήθελα να γνωρίζω όμως είναι ποια ήταν η εμπειρία σας στην, ε, όσον αφορά αυτή την πρόκληση και επίσης ε, σε σχέση με την αρχή της ανεξαρτησίας των κρατών μελών ε, ε, ως προς αυτό το θέμα και τι θα πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης, τι ε, συμβουλή θα δώσετε στον ή στην διάδοχό σας ώστε να ε, ε, ε, βελτιωθεί η κατάσταση του ανθρώπου που υφίσταται τα χειρότερα διακρίσεις στην Ευρώπη, δηλαδή την γυναίκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ξέραμε ότι θα πυροδοτούσατε την προσοχή όλων στην ε, Επιτροπή μας, νέων και παλαιών ε, βουλευτών. Πολύ ζεστή συζήτηση, πολύ ζωντανή. Ε, παρακαλώ λοιπόν τώρα να κάνετε ό,τι μπορείτε να δώσετε τις απαντήσεις και θυμίζω πως υπάρχει πάντοτε δυνατότητα κάποιες διευκρινήσεις να δοθούν γραπτός στη συνέχεια για όσους πέβαλαν πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι καλό να μπορέσω να απαντήσω και γραπτός, γιατί δεν ισχυρίζομαι ότι τα ξέρω όλα. Κάποιες ερωτήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες γιατί είχαν και κάποια νομική φύση ε, και απαιτείται κάποια ακριβής ε, διατύπωση, οπότε μπορείτε να μαζέψετε όλες μαζί τις ερωτήσεις που δεν θα απαντήσω και να μου τις ε, στείλετε, θα απαντήσουμε. Θα ξεκινήσω από το τέλος την ερώτηση για το φύλλο. Είχαμε μια στρατηγική η οποία καλύπτε πολλές προτεραιότητες. Η πρόοδος ε, δεν είναι μεγάλη, λυπούμε. Πρέπει να πω ότι σε κάποιους από τους δείκτες π.χ. απασχόληση, το μισολογικό κενό, ε, γυναίκες ε, στα θεσμικά όργανα ανεβαίνει σιγά σιγά αλλά δεν είναι κάτι το εκπληκτικό. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 36% στο 40% είναι κάποια πρόοδος. Αλλά η Συμβουλή για τις γυναίκες πολιτικούς είναι εξής. ακούσαμε χθες την Τερέζα Μέη ε, είπε χθε στη Βουλή να είστε ο εαυτός σας. Ε, εντάξει, δεν πρωτότυπο, αλλά μου άρεσε αυτά τα οποία είπε χθε το δεύτερο για να ξεκαθαρίσει μία παρεξήγηση όταν είπα ότι ε, το κράτος δικαίου ε, ε είναι εμπόδιο. Προφανώς ε, δεν είπα κάτι τέτοιο. Το εννοούσα το εξής. Όταν είπαμε συγχωρείτε ότι είναι κάτι το αφηρημένο. Να είναι ότι δεν είναι μετρήσιμο αυτό το οποίο εννοούσα. Και το δεύτερο, πίστεψτε με, δεν είναι εύκολο και το ξέρετε ε, να εξηγήσουμε στους ε, πολίτες ε, που δεν είναι δικηγόροι και δεν έχουν μελετήσει το συνταγματικό δίκαιο γιατί είναι τόσο σημαντικό. Γιατί είναι τόσο σημαντική η αρχή ότι ο νικητής των εκλογών δεν παίρνει τα πάντα είναι μια αρχή στην οποία βασίζονται οι δημοκρατικές κοινωνίες και παραδόξως ε, δεν καταφέρνω να το εξηγήσω σε πολλούς γιατί είναι τόσο σημαντικό. Ίσως να είναι θέμα επικοινωνίας, πρέπει να τα πάμε καλύτερα και να σκεφτούμε ίσως ε, την εκπαίδευση για τις βασικές αρχές ε, των δημοκρατικών κοινωνιών. Τρίτον, Για, λέτε ότι ε, απάντησα με κάποια προκατάληψη. Όχι, όχι, δεν. Απάντησα αυτά τα οποία πρόλαβα και μου αρέσουν οι δύσκολες ερωτήσεις. Ε, γιατί ακριβώς ε, είναι δύσκολα ζητήματα αυτά και τα ζητήματα ταυτότητας. Συνήθως δεν υπάρχει η θέληση να γίνουν συμβασμοί. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα για να απαντώ και σε δυσάρεστες ερωτήσεις. Ε, λοιπόν, θα επανέλθω ε, στην κυρία Ρέιτ και γιατί ρώτησε κάτι για το κράτος δικαίου σε σχέση με τον προπολογισμό. Ελπίζω να εγκριθεί και η πρόταση για την σχέση μεταξύ κράτους δικαίου και προπολογισμού είναι πολύ συγκεκριμένη. Η διαδικασία η οποία προβλέπεται είναι πολύ ισορροπημένη, οπότε θεωρώ ότι θα περάσει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και επίσης το ζήτημα για την οικογενειακή βία κατά γυναικών και παιδιών. Βασιζόμαστε στο ότι θα κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη και στην βεβαιότητα του ότι θα συνυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό της αρμοδιότητάς της. Ε, τίποτα από αυτά δεν συνέβη όμως δεν είναι επιτυχία. Και ειλικρινά προσπάθησα πάρα πολύ να γίνει αυτό. Βεβαίως ε, η κύρωση της συνθήκης είναι κυρίαρχο δικαίωμα των κρατών μελών, οπότε πρέπει να το σεβαστώ αυτό. Βεβαίως προσπάθησα να εξηγήσω και σε κάποιες χώρες γιατί η σύμβαση αυτή ε, θεωρείται χρήσιμη χωρίς την σύμβαση αυτή για το μέλλον, ίσως τα πράγματα θα είναι χειρότερα. όσον αφορά κάποια συγκεκριμένα νομοθεσία για κάποια συγκεκριμένα εγκλήματα. Η κυρία Πρόεδρος είπε επίσης ότι θέλει να κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά γνωρίζετε πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα του ποινικού δικαίου πάντα υπάρχει ε, μια διαμάχη, αν θέλετε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών για το τι πρέπει να ρυθμιστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε είναι χειρότερα τα πράγματα για κάποια νομοθετήματα γιατί η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν θα έχει τόσο εύκολο μέλλον μετά. Για τον πίνακα βαθμολογίας ε, και θα αναφερθώ και στο μηχανισμό CVM ε, και την βαθμολογία εκεί. Έχουμε πολλά μέσα για να εξετάζουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη. Έχουμε το άρθρο 7 που είναι η τελευταία λύση όταν βλέπουμε συστημική παραβίαση του κράτους ε, δικαίου. Έχουμε τον πίνακα βαθμολογίας. Κάποιοι το ρωτήσατε. Το θεωρούμε ένα πολύ χρήσιμο μέσο που μετράμε την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα και κάποιους άλλους μετρήσιμους δείκτες για την δικαιοσύνη και κάποιες ε, δείκτες αξιών όπως η ανεξαρτησία και η ποιότητα της δικαιοσύνης. Κάθε χρόνο βεβαίως αυτό συγχύζει κάποιους υπουργούς δικαιοσύνης ε, ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση της αντίληψης των πολιτών και των επιχειρήσεων που είναι πάντα ένα ευαίσθητο θέμα. υπάρχει κάποιο συσχετισμός μεταξύ τη χαμηλή εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη και του πόσο εύκολα μπορούν να επιτεθούν οι πολιτικοί στην δικαιοσύνη. Όταν είναι χαμηλή η εμπιστοσύνη των πολιτών, δεν κοστίζει τίποτα στον πολιτικό να επιτεθεί στην δικαιοσύνη, γιατί ο λαός είναι μαζί σου. Δεν το βλέπω αυτό σε πολλά κράτη-μέλη. Οι επιθέσεις κατά της δικαιοσύνη είναι δημοφιλείς ε, σε κάποια κόμματα της κοινωνίας. Για πρέπει να προσέχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, ο πίνακας βαθμολογίας. Θα συνεχίσουμε, θα θέλαμε να έχουμε και άλλα κεφάλαια, ειδικά που θα αφορούν το ποινικό δίκαιο. Μετά. Το τρίτο σύστημα είναι η στάση αναχώρα που χρησιμοποιούμε. Γιατί, γιατί αυτό αφορά την οικονομία. Αλλά βεβαίως και η λειτουργία της δικαιοσύνης επηρεάζει πολύ τις οικονομικές συνθήκες μιας χώρας. Τα έχουμε αυτό το οποίο προτάθηκε, μια ετήσια έκθεση για το κάτω δικαίου και έχουμε και τις ειδικέ εκθέσεις για δύο χώρες, Βουλγαρία και Ρωμανία και θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ότι ο μηχανισμός για τις δύο αυτές χώρες πρέπει να τελειώσει ε, όταν οι χώρες οριστικοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις και ακολουθήσουν τις συστάσεις. Είναι κάτι το οποίο ε, είναι αντικείμενο εντατική συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κρατών Μελών. Προσωπικά έχω μιλήσει πολλέ φορέ με του Υπουργού Δικαιοσύνη, ε, του εισαγγελεί για το πώ μπορεί να βοηθήσει η Κομισιόν Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν ε, και τα πράγματα είναι αυτά τα οποία ε, ίσχυαν και τον Οκτώβριο του 2018. Αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω την δήλωση Γιούνκερ. Και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Τώρα, γιατί υπάρχει ειδική μεταχείριση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ήταν ε, κάτι το οποίο είχε συμφωνηθεί με την ένταξη των χωρών αυτών και πρέπει να οριστικοποιηθεί με κάποια πραγματική ε, πρόοδο και αποτελέσματα. Νομίζω είναι προς το συμφέρον και των χωρών αυτών και της Κομισιόν. Το θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που επίσης σχετίζεται με το κράτος δικαίου. Έχουμε πολλά μέσα που σχετίζονται με αυτό το ευρωπαϊκό ένταλμα τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Υπήρχε ένα ερώτημα σχετικά όταν συζητήσαμε τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία στο Συμβούλιο. Υπάρχουν δύο ζητήματα. Σεβασμός ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, σεβασμός εξαρτωμένων μελών ε, και ατόμων ε, των οποίων τα δεδομένα χρησιμοποιούνται σε μια έρευνα και βεβαίως η εμπλοκή των εταιριών πληροφορικής σε μια άλλη χώρα. Ε, για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν μου αρέσει το πώς λειτουργεί τώρα, γιατί τώρα ε, ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει τα δεδομένα και μπορεί να το κάνουν είτε όχι, είναι θελοντικό. Ανάλογα με το αν κοιμήθηκε καλά ο διευθύντης, εντάξει υπερβάλλω, αλλά δεν έχει κάποια αξιοπιστία η διαδικασία. Είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και γνωρίζουμε ότι ο μηχανισμό αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει μια ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι το οποίο δεν ισχύει αυτή τη στιγμή γιατί υπήρχαν κάποιε πολύ έντονε συζητήσει. Επίση, όταν πηγαίνω στη ΣΥΠΑ και μιλάμε για μια ευρωπαϊκή συμφωνία με τη ΣΥΠΑ και ακούω ότι οι ΙΠΑ θα επιλέξουν κάποιες χώρες. Πρέπει να πω όχι. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουμε κοινέ προδιαγραφέ. Αλλά πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, πηδά από το ένα στο άλλο. Γιατί νιώθω εδώ πέρα ότι κάτι θέλετε. Όχι, όχι, λέει ο πρόεδρο, μην ανησυχείτε. Είναι ε, μια χαρά, δεν μην νιώθετε τίποτα. Όχι, ε, πόσο χρόνο έχουμε όμω. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μα, εντάξει, προφανώ. Αλλά θα ζητήσουμε συγγνώμη από την επόμενη παρουσίαση που είναι ακριβώ ο πίνακας βαθμολογίας ε, που σχετίζεται με αυτά τα οποία μας λέτε. Το κάλυψε αυτό. Βεβαίω ε, για την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα μέσα. Υπάρχει ε, η σοβαρή νομολογία του δικαστηρίου που λέει ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση υψηλών προτεγραφών παντού και να πάρουμε σοβαρά όλα αυτά τα ευρήματα και τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν περισσότερα. Τέλος, έχουμε την τελική συμφωνία μεταξύ ε, ΕΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Ε, η κυρία Νετφελτ νομίζω ήθελε να πάει στο ΔΕΚ για να κρυθεί. Αυτό είναι το νομικό θέμα που πρέπει να εξετάσουμε αλλά εντάξει δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. CVMI. Πήγα να το καλύψω μετά. Κράτηση και ζητήματα ισότητας, κύριε Παγκάζα... Βουντούα Μάλιστα. Α, πρέπει να τα μάθω. Έμα, ε, όνομα είναι αυτό, λέει ο πρόεδρος. Βεβαίως ε, η κράτηση και τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι μεγάλο θέμα και πρέπει ακριβώ τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στις απαιτήσει ε, του ΕΔΑΔ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε μια μακροσκελή συζήτηση με τους υπουργού για τις συνθήκες κράτησης, εναλλακτικέ ποινές, ε, τους πρώτους να χρησιμοποιήσουν περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, τώρα δεν έχουμε χρόνο, αλλά είπα συγκεκριμένα του που βρίσκονται τα λεφτά. Και πάλι, ε, για να είμαι κάπως ειλικρινής, μου λένε τα κράτη-μέλη ότι δεν ε, είναι πολύ δημοφιλές να επενδύουν σε φυλακές. Ε, ότι θέλει ο κόσμος να επενδύουν σε σχολεία και νοσοκομεία. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι και εγώ είμαι πολιτικός, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν σεβαστά έχουμε κάποιες ε, δυνατότητες να συνεισφέρουμε από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να αυξηθεί το επίπεδο στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για να επανέλθω λίγο στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και την ανταλλαγή δεδομένων. Έχουμε τώρα τρία μέσα που χρησιμοποιούμε στο ποινικό δίκαιο. Η αμοιβαία συνδρομή όταν ο δικαστή ε, ζητά ε, συνεργασία. Χρειάζονται 10 μήνε κατά μέσο όρο για να λάβει μια απάντηση. Όταν χρησιμοποιούν ε, το Ευρωπαϊκό Εντέλμα έρευνα 120 μέρες. Τώρα προσφέρουμε ένα σύστημα με τις απαραίτητες δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιώματα των υπόπτων και των θυμάτων και των μαρτύρων ή να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα, προσφέρουμε ένα μέσο το οποίο σε κρίσιμες στιγμές θα επιτρέψει στις διοκτικές αρχές να, ε, να δώσουν τα αποδεικτικά στοιχεία σε 7 ώρες ή σε 10 μέρες. Ε, μιλάμε για επανάσταση. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό χρειάστηκε τόσο καιρό για την Κομισιόν για να προετοιμάσει αυτή την πρόταση, γιατί το δουλεύαμε δύο χρόνια, ήρθαμε τον Απρίλιο πέρσι. Εντάξει, αργά το παραδέχομαι, αλλά θέλαμε να το κάνουμε σωστά. Και είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε περισσότερες δικλείδες ασφαλείας, πιο έντονη εμπλοκή του κράτους μέλους που ζητάει την επιβολή κτλ. Οτιδήποτε απαιτείται. Κύριε Ενσέρα, για την υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα εγκλήματα που αφορούν τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, συλλέγουμε τα δεδομένα. Υπάρχει διαδικασία παραβάση κατά πολλών κρατών μελών για έλλειψη εφαρμογής ε, του πλαισίου για ρατσισμό, ξενοφοβία κτλ. Το εάν ε, η Κομισιόν θα προτείνει να διευρυνθεί και σε Άλλες ομάδες ε, πολιτών ε, όχι ακόμα, όχι. Ίσως η επόμενη επιτροπή. Για την οδηγία ε, περισσότητας, όπως είπα, πρέπει να προσπαθήσουμε ξανά. Η επόμενη ευκαιρία μας είναι τον Οκτώβριο. και Κενερικό, συνεργαζόμαστε με όσα και άλλους οργανισμούς για το ξεπλήμα χρήματος. Βεβαίως, συνεργαζόμαστε πρώτα απ' όλα στο πλαίσιο αυτής της ε, Task Force που είναι βασική, ο βασικός οργανισμός. Όμως, αποφασίσαμε να κάνουμε περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό κάνουμε. Η νομοθεσία Ε, για την τέταρτη και πέμπτη οδηγία, ε, για την εφαρμογή τους και για δράσεις στον πραγματικό κόσμο. Πώς είναι δυνατόν στην Εστονία, σε ένα υποκατάστημα της Danske και Bank να ξεπλύνουν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε 7 χρόνια. Δεν το πρόσεξε κανείς. Μιλάμε για ε, κανόνες ντοσχέ ολόκληρα. Τσεκάρουν τα κουτάκια υποτίθεται και υπάρχει εποπτεία. Ε, και όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πώς είναι δυνατόν. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε κάποιες απαντήσεις ε, και είχαμε κάποιες και πολύ συγκεκριμένα διδάγματα από την περίπτωση αυτή. Στην ε, χθεσινή έκθεση της Κομισιόν, ε, δείτε το. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Οι νέες τάσεις, οι ελευθερλημένες, ανώνυμες συναλλαγές, ε, πώληση υπηκοτήτων. Πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα. Αν μου επιτρέπετε λέει πρόεδρος. Ναι, δύσκολα είναι. Έτσι είναι. Πάντα στην Επιτροπή μας ο χρόνος πιέζει. Ε, σας παρακαλώ να, να συντομεύετε. Λοιπόν, ε, το ε, ψηφιακό νόμο είναι άλλη γενική διεύθυνση. Δεν ξέρω τι σχεδιάζουν. Έχω ένα όραμα δικό μου εγώ, αλλά δεν θέλω τώρα να σας ε, μπερδέψω και σας και άλλους για να βγουν να πούνε ότι η Γιούροβα δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και μπρος και λέει διάφορα. Είναι άλλη γενική διεύθυνση. Κύριε Σδεχόφσκι, το μεγαλύτερο πρόστιμο για την Cambridge Analytica ήταν μισό εκατομμύριο λίρες στη Μεγάλη Βρετανία. Συνεχίζονται οι έρευνες, αλλά η κατάσταση και το τόσο χαμηλό ε, πρόστιμο δείχνει πως ακριβώς ο κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων ε, χρειαζόταν, που έχει υψηλά πρόστιμα και ε, στην περίπτωση αυτή πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες που ίσχυαν πιο πριν βεβαίως και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τι άλλο. Ε, διπλά διτά προϊόντα είναι θέμα προστασίας καταναλωτών, μεγάλη υπόθεση πρέπει να συνεχιστεί. Η νομοθεσία είναι ένα ε, προϊόν συμβασμού δηλαδή απαγορεύεται η διτυπιότητα εκτός εάν υπάρχει κάποιος ε, σοβαρός λόγος, παραδείγματος χάρη εθνικές προδιαγραφές που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οπότε ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά η Κομισιόν προετοίμασε την μεθοδολογία για τις δοκιμές ε, τροφίμων έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στις εθνικές αρχές ε, για επιθεωρήσεις και ήδη έχουμε εκδώσει νομική γνωμοδότηση ότι πρόκειται για την εμπορική πρακτική και μπορεί να τιμωρηθεί τώρα επαφίεται στις ε, επιθεωρήσεις των κρατών μελών. Έχω συνεχή συζήτηση με τους παραγωγούς, έχω κατονομάσει εταιρείε ε, τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε την συνεχή συζήτηση με τις βιομηχανίες τροφίμων. Πιέζω όσο μπορώ, αλλά τώρα πρέπει να τα δουν αυτά οι εθνικές επιθεωρήσεις. Από τον Ιανουάριο του 20 θα υπάρχει ο νέος κανονισμός για καλύτερη συνεργασία των ε, επιθεωρήσεων ε, τροφίμων διασυνοριακά μπορούν να δημιουργήσουν κοινά δίκτυα και να κυνηγήσουν την υπόθεση. Αυτά σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε εμείς πολύ κύριε Επίτροπε και εκτιμούμε πολύ τις προσπάθειές σας και βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και περιορισμοί χρόνου. Ευχαριστούμε που παρατείνατε τον χρόνο που μας αφιερώσατε, παρόλο που η επίσκεψη σήμερα... Όσοι εξημών θέσατε ερωτήσεις σχετικά με την ε, δικανική συνεργασία για ποινικά θέματα. Υπάρχει περιθώριο να συζητηθεί το θέμα αυτό και στο επόμενο ζήτημα της ημερήσιας διάταξης που είναι η εξέταση του βαθμολογίου της δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ανακοινώνω ότι η υπόλοιποι Επίτροπη που έχουν ειδικά χαρτοφυλάκια αρμοδιότητα τη Επιτροπή μα αρχέ Σεπτεμβρίου, δηλαδή τον Αντιπρόεδρο κ. Τίμερμαν για ανθρώπινα δικαιώματα στι 4 και 5 Σεπτεμβρίου και τον κύριο Αβραμόπουλο, αρμόδιο για εσωτερικά, στις 12 Σεπτεμβρίου. Προχωρούμε τώρα στο βαθμολόγιο της δικαιοσύνης, Justice Scoreboard. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Επίτροπο και της ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.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 Χωρίς άλλες καθυστερήσεις να πάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης που, ε, για το οποίο προβλέπονται 45 λεπτά βέβαια αλλά ίσως μπορέσουμε να συντομεύσουμε για να έχουμε λίγο χρόνο και για το επόμενο, δηλαδή το μεθ επόμενο θέμα. Έχουμε κάτι που ακόμα δηλαδή στην ημερησία διάταξη. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την εξέταση όπως είπα και πριν του ε, βαθμολογίου δικαιοσύνης. Όσοι δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό το πράγμα, υποτίθεται ότι είναι ένα συγκριτικός μηχανισμός πληροφόρησης στην βάση διαφόρων δικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας, ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας των δικανικών συστημάτων ε, σε όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης. Οι βασικές παράμετροι είναι οι εξής τρεις ανεξαρτησία, ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί ήδη από το 2013 και μέχρι το 2019 έχουν προσθεθεί και άλλοι δείκτες επικοινωνία και ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχόμενα νέα βήματα. Αυτά εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2019 μέσα σε αυτό το ε, βαθμολόγιο που θα είναι και ένα νέο μηχανισμό για την ενίσχυση του κράτου δικαίου, για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη και των προτύπων κράτου δικαίου. Μας απασχολούν ιδιω αυτή η σταδιακή μείωση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων δικαστηρίων, δηλαδή τα οποία ωστόσο περιλαμβάνονται στην Συνθήκη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θεωρούμε σωστό πριν από την ε, θερινή διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου <clears throat> να το συζητήσουμε και σας δείχνω εδώ και το σχετικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε. Έξω στα τραπέζια, έξω από την αίθουσα της ε, Επιτροπής ε, Θεμελιδών Ελευθεριών, ο κύριος Ντέλ της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι παρόν το άτομο αυτό. Μάλιστα, ορίστε. Έχετε το λόγο κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να σας ενημερώσουμε για την έκδοση 2019 του ε, βαθμολογίου το οποίο εξετάζει αριθμό δικτών της ανεξαρτησίας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εθνικών δικανικών συστημάτων. Για το 2019, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο, αυτή ήταν η έβδομη έκθεση, και μέσα στα χρόνια ε, ο μηχανισμός αυτός έχει εξελιχθεί και είναι σημαντικός μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Ακούσαμε πριν από την Επίτροπο κυρία Γιούροβα ε, σχετικά με τους τρόπους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει το ε, βαθμολόγιο. Και αυτά περιλαμβάνονται και στι ανακοινώσει τη προηγούμενη εβδομάδα που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και βεβαίω και περαιτέρω εξέλιξη του βαθμολογίου. Και θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Από την πρώτη έκδοση του 2013, το Justice Scoreboard έχει ήδη εξελιχθεί σημαντικά. Η πρόοδος οφείλεται και στις εισρωές της παρούσας Επιτροπής και την ενθάρρυνσή της και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γενικότερα, το οποίο έχει ε, ψηφίσει τρία ψηφίσματα για το βαθμολόγιο τα τελευταία χρόνια. Στόχος του βαθμολογίου είναι να ε, συμβάλλει στην ε, βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δικανικών συστημάτων των χωρών μελών. Το βαθμολόγιο δεν προχωρεί σε ιεράρχηση, προσφέρει συγκρίσιμη αξιόπιστη πληροφόρηση για τη λειτουργία των δικανικών συστημάτων, των συστημάτων δικαιοσύνη δηλαδή, που υποτίθεται ότι οδηγούν και σε περαιτέρω βαθύτερε σκέψει για του λόγου που προκύπτουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Και γίνεται και βαθύτερε αξιολογήσει αναχώρα σε διμερή διάλογο με τι εθνικέ αρχέ και συμφεροντούχου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και επιτρέπουν έτσι να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των δικανικών συστημάτων των χωρών μελών, η ανεξαρτησία, ποιότητα και αποτελεσματικότητα λοιπόν, που είναι τα τρία στοιχεία ενώ για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα δικαιοσύνης, είναι σημαντικά για τη διατήρηση του κράτου δικαίου. Αποτελεσματικά δικανικά συστήματα είναι επίση σημαντικά για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί τα εθνικά δικαστήρια ε, ενδύονται το μανδύα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όταν εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και έχουν σημαντική ε, πυροή έτσι και στα επενδυτικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα των χωρών μελών και άρα στην οικονομική τους ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς το Justice Scoreboard ε, τροφοδοτεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με τις ειδικές εκθέσεις αναχώρα και τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Όπω είπαμε και στην ανακοίνωση της προηγούμενη εβδομάδα το βαθμολόγιο θα τροφοδοτεί και τις μελλοντικέ αιτήσει εκθέσεις κράτους δικαίου, τις οποίε θα συντάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα στην 7η χρονιά που εκδίδεται το Justice Scoreboard και βλέπουμε ήδη να διαγράφονται κάποιες τάσει. Τα αποτελέσματα του φετινού χρόνου είναι μεικτά, ανάμεικτα. Δείχνουν σχετικές βελτιώσεις ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των ε, συστημάτων απονομής δικαιοσύνης σε πολλές χώρες, αλλά δυστυχώς σε ορισμένες χώρες οι τάσεις αναστρέφονται και η κατάσταση επιδεινώνεται. Στα πλαίσια αυτά, το χαμηλό επίπεδο της αίσθηση που έχουν οι, οι πολίτες για την ε, απονομή δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Να αρχίσω όμως με τις θετικές τάσεις. Τα τελευταία 8 χρόνια είδαμε μια συνολική θετική ε, τάση αύξησης της αποτελεσματικότητας των δικαστηρίων. Η διάρκεια των ε, δικαστικών διαδικασιών στο αστικό δίκαιο έχει μειωθεί ή πάντως έχει παραμείνει σταθερή. Και το ίδιο ισχύει και τι περισσότερες χώρες μέλη και σε ό,τι αφορά τις διοικητικέ υποθέσεις που δικάζονται. Παραδείγματα, υπάρχουν χώρες οι οποίες μείωσαν σημαντικά την διάρκεια των διαδικασιών μεταξύ 2010 και 2017, καθώς και τις καθυστερούμενες υποθέσεις, για παράδειγμα Σλοβενία, Σλοβακία, Κροατία, Παίρνοντα κανεί όλε τι υποθέσει αστικού δικαίου, η Κροατία μείωσε τι καθυστερούμενε υποθέσει κατά 30%, η δε Σλοβενία κατά 70%. Η διαδικασία, μάλλον το, η διάρκεια των διαδικασιών έχει μειωθεί και στην Ιταλία, παραμένουν όμω σημαντικέ προκλήσεις και ιδίως στου υψηλότερου βαθμούς απονομή δικαιοσύνη. Εκτός από την ε, αποτελεσματικότητα, εξετάζει το βαθμολόγιο και την ποιότητα. Οι περισσότερες χώρες μέλη διαθέτουν προδιαγραφές για την ε, ενημέρωση των διαδίκων για ενδεχόμενες καθυστερήσεις, για την πρόοδο διαδικασίας. Έχουν επίσης βελτιώσει την επιγραμμική πρόσβαση ε, στις υποθέσεις και ιδίως στις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, 19 χώρες μέλη δημοσιεύουν όλες τις ε, εμπορικές και αστικές αποφάσεις. Ο προϋπολογισμός, οι προϋπολογισμοί μάλλον της δικαιοσύνης παραμένουν σταθεροί, μάλιστα ένας αριθμός χωρών μελών έχουν αυξήσει τον προϋπολογισμό για τη δικαιοσύνη και αναφέρω εδώ την Ιρλανδία, Φιλανδία και Λετωνία Για πρώτη φορά επίσης έχουμε βελτίωση ε, της ποιότητας των αποφάσεων. Βλέπουμε σε ένα αριθμό χωρών μελών να υπάρχουν μηχανισμοί πλέον για τη διευκρίνηση των αποφάσεων και την τάση να χρησιμοποιούν απλή, ξεκάθαρη γλώσσα. Βλέπουμε επίσης ότι τα δικανικά συστήματα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες συγκεκριμένων διαδίκων όπως παιδιών και την ίδια έκδοση υπάρχει και ένα νέο κεφάλαιο που αναφέρεται στις ε, ε, κρατικές δαπάνες για τα δικαστήρια. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πρέπει να υπάρχει μια κοινή κατανόηση ότι οι επενδύσεις στη δικαιοσύνη θα αποτελούν κόστος. Αντιθέτως, όταν στοχεύονται καλά οι επενδύσεις αυτές, αποτελούν πραγματικές επενδύσεις. Να έρθω τώρα στα καινοτόμα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία. Για πρώτη φορά έχουμε δημοσιεύσει επισκόπηση των αρχών που εμπλέκονται σε επιθαρχικές διώξεις δικαστών, οι οποίοι δικαστές οφείλουν να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να ε, λαμβάνουν αποφάσεις στις υποθέσεις που δικάζουν χωρίς κανένα επηρεασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφύγει κατά της Πολωνίας για να αποφευθεί η προσπάθεια επηρεασμού δικαστών. Και έχει εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη και έχει δώσει δύο μήνες προθεσμία στην πολωνική κυβέρνηση για να απαντήσει. Όπως θα δείτε στο βαθμολόγιο, οι λύσεις που προτείνει η Πολωνική Βουλή περιλαμβάνει και, περιλαμβάνουν και ε, καινοτόμα στοιχεία, μοναδικού χαρακτήρα. Ερχόμαστε τώρα στις βασικές προκλήσεις που ε, αναφύονται μέσα από το ε, βαθμολόγιο. Πρώτα, οι χώρε μέλη οφείλουν να πράξουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τι καθυστερούμενε υποθέσει και να μειώσουν τη διάρκεια των διαδικασιών και ιδίω στι χώρε οι οποίε έχουν εντοπιστεί και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ότι αντιμετωπίζουν δηλαδή, τι μεγαλύτερες προκλήσεις. Τον Ιούλιο, το Συμβούλιο μετά από πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απίφθινε ειδικέ συστάσει σε 7 χώρε μέλη. Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Ουγγαρία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβακία. Δεύτερο λοιπόν, τώρα υπάρχει χώρος βελτίωσης και για την χρήση και πρόσβαση σε ηλεκτρονικά εργαλεία, για την παρακολούθηση ας πούμε ε, δικαστικών διαδικασιών επιγραμμικά. Τονίζω επίσης ότι η ανεξαρτησία δικαστηρίων και δικαστών παραμένει ένα θέμα σε ορισμένες χώρες μέλη και συστάσεις ειδικέ αναχώρα για τρεις χώρες αναφέρονται ακριβώς αυτό το θέμα. Εξετάζοντας τώρα το βαθμολόγιο του 2019, βλέπουμε ότι οι παρεμβάσεις και πιέσεις πολιτικών προσώπων είναι ο βασικός λόγος στα μάτια πολιτών και επιχειρήσεων για να θεωρήσουν ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. 7 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η δικαιοσύνη δεν είναι ασφαλής ιδίω λόγω παρεμβάσεων και πιέσεων πολιτικών. Και αυτό δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει να είναι ασφαλές το δικαστικό σύστημα απέναντι σε τέτοιες παρεμβάσεις. Και για να είμαι σαφής, ήδη λέχθηκε προηγουμένω από την Επίτροπο κ. Γιούροβα ότι εάν ένα σύστημα απονομή δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σωστά σε μία χώρα μέλο, οι επιπτώσει θα γίνουν αισθητέ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αμοιβαία εμπιστοσύνη οι αποφάσεις δικαστηρίων μιας χώρας αναγνωρίζονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να υπάρχει σκιά αμφιβολίας για την ανεξαρτησία των δικαστών που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την νέα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω εξέδωσε την ανακοίνωση. Όπως δηλώνει η ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσπαθήσει να βελτιώσει και το ίδιο το βαθμολόγιο, ώστε να καλύπτει και άλλα θέματα κράτου δικαίου και ιδίως στον τομέα της ποινική δικαιοσύνης. Και αναμένουμε τις εισρωέ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτές και ιδίω από την παρούσα Επιτροπή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντέλ για την παρουσίαση του θέματος που συνδέεται ασφαλώς με την συζήτηση που διεξήχθη μόλις πριν με την Επίτροπο κυρία Γιούροβα. Ασφαλώς λοιπόν αναμένω κάποιες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις μετά από τις ανησυχίες που ακούστηκαν προηγουμένως στο πρώτο τμήμα της συνεδριασής μας. Αρχίζουμε με τον κύριο Ζαβόσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι είμαι ο μέγας σπεσιαλίστας ε, της διαδικασίας του βαθμολογίου. Τέλος πάντων, ε, για να είμαι πιο σοβαρός τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία που κάνετε και έχετε κάνει πολλά πράγματα, αλλά βλέπω να μου λείπουν πολλές πληροφορίες από πολλές χώρες. Επίσης, πώς μπορείτε να συγκρίνετε το γαλλικό σύστημα με το τσεχικό. Πώς μπορείτε να συγκρίνετε την ποιότητα της απονομής δικαιοσύνης σε κάθε χώρα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορώ να σα εξηγήσω στο τσεχικό σύστημα που εξακολουθούν να μην λειτουργούν. Και είμαστε πλέον στον 21ο αιώνα. Εξετάστε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Πόσες χώρες έχουν ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Πόσες χώρες χρησιμοποιούν ψηφιακές μεθόδους για την ε, παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ε, ε, εργασιών των δικαστηρίων. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε πολλά νούμερα, μπορούμε να τα εξετάσουμε, αλλά δεν μας επιτρέπει αυτό να κρίνουμε ποιοι τα πάνε καλά και ποιοι όχι. Υπάρχουν και πολλές μεθοδολογικές αλλαγές που μπορεί να δει κανεί μέσα στον χρόνο. Ακόμα δεν έχουμε όμως μία ενιαία μεθοδολογία για να συγκρίνουμε τα συστήματα μεταξύ των χωρών. Και σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα της δικαιοσύνης και την ουδετερότητα των δικαστηρίων και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πολλά πράγματα τα ακούμε από τον τύπο. Κανείς όμως δεν μπορεί να πει πραγματικά και ουδέτερα κάτι τι για την ποιότητα των δικαστηρίων εάν βρίσκεται εκτός του συστήματος. Και τώρα για το για τα πολιτικά συμφέροντα σε πολλές υποθέσεις. Είχαμε ένα πρωθυπουργό που είχε τεράστιο πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων και τώρα ανακρίνεται από την αστυνομία και όμως εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. Ε, πώς μπορείτε να πείτε τώρα κάτι για την δικαιοσύνη στην τσεχική δημοκρατία, εάν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό της χώρας που ασκεί την εξουσία επικρίνει το έργο της αστυνομίας, επικρίνει το έργο της δικαιοσύνης, αλλάζει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, διότι υπήρχε το πρόβλημα ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριζε την ε, ουδετερότητα των ανακρίσεων. Δεν θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα ε, στο βαθμολόγιο. Να με συμπαθάτε που μακρηγορώ, αλλά είναι κρίμα γιατί κάνετε πολλή δουλειά και σας ευχαριστώ για την πολλή δουλειά που κάνετε, αλλά τα αποτελέσματα για μένα ε, είναι στην πραγματικότητα τίποτα, μηδενικά. Λυπάμαι πολύ που χρόνο να πω αυτά. Πρόεδρος Αγγιλάρη, μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Και μην λησμονείτε επίση, βεβαίως όλες οι παρεμβάσει είναι καλοδιχούμενες αλλά το βαθμολόγιο δικαιοσύνη δημιουργήθηκε ακριβώς μετά από αίτημα της Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε που ήταν επίτροπος η Vivian Redding Βεβαίως και γνωρίζαμε ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία και ανομοιογένεια ανάμεσα στα δικανικά συστήματα των 28 χωρών μελών και ότι είναι διαφορετικός ο χαρακτήρας των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και ακριβώς ένα εργαλείο που να επιτρέπει τη σύγκριση, τη συγκριτική ανάλυση είναι ένας τρόπος να γίνει πιο αντικειμενική η, ε, ε η ενατένιση του που βρίσκεται πως ε, αποδίδει το κάθε σύστημα. Όπως είπα, ε, ποιότητα, ανεξαρτησία και αποτελεσματικότητα. Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω την ε, Κομισιόν για την παρουσίαση που έκανε για τα δεδομένα του πίνακα βαθμολογίας. Βεβαίω είναι σημαντικό να έχουμε δεδομένα συγκρίσιμα για να γνωρίζουμε την κατάσταση της δικαιοσύνης ε, σε όρους αποτελεσματικότητας ε, και ποιότητας. Αλλά και εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Θα ήθελα συγκεκριμένα να αφαιρθώ στο θέμα της ανεξαρτησίας της ε, δικαιοσύνης που είναι ένα θέμα λεπτό και περίπλοκο. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Με ποιον τρόπο το μέσο αυτό του πίνακα βαθμολογίας μπορεί να συνεισφέρει συγκεκριμένα στο να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στα κράτη-μέλη. Και άλλη μια ερώτηση κάπως πιο συγκεκριμένη σε σχέση με τα δεδομένα για τις διώξεις, για το ξέπλυμα χρήματος ε, που προκύπτουν εδώ από την ανάλυση του πίνακα βαθμολογίας. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν εάν έχει σήμερα, γιατί το θέμα του ψεπλήματος ε, το είδαμε πριν και με την κυρία Γιούροβα, είναι πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω λοιπόν εάν σήμερα έχει δεδομένα για την πλήρη διάρκεια των διαδικασιών αυτών στις ε, χώρες ε, και για το τι γίνεται με τις καταδίκες και Θα ήθελα να ρωτήσω αν η Κομισιόν σκοπεύει σε μια επόμενη έκδοση να περιλάβει τέτοια στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Κυρία Στρίκ ε, για τους πράσινους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την ε, παρουσίασή σας αυτή. Έχω δύο σύντομες ε, ερωτήσεις. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με τις προτάσεις ενίσχυσης του συστήματος, αλλά αναρωτιόμασταν αν οι δείκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή επαρκούν για να μετρήσουμε το επίπεδο ποιότητας του κράτους δικαίου και είναι λίγο πολύ ποιοτική σε πολλές περιπτώσεις, αφορούν και τη διάρκεια της διαδικασίας ή ε, είναι περιορισμένοι στις διαδικασίες που περιγράφονται στα χαρτιά ενώ εάν θέλουμε να δούμε το επίπεδο ανεξαρτησίας και ποιότητας, πρέπει να δούμε και το τι γίνεται στην πράξη και ίσως την ποιότητα των αποφάσεων. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν εάν χρειάζονται και άλλοι δείκτες και αν είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Και το άλλο. Θα μπορούσε ο πίνακας βαθμολογίας να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ε, υπάρχει τώρα η σχέση με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα μπορούσε να συνδεθεί και με τη χρηματοδότηση της Ένωσης και γνωρίζω πως υπάρχει αυτός ο κανονισμός για... Πώς λέγεται... Που εκκρεμεί τώρα σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για να συνδεθεί με την κοινοτική χρηματοδότηση Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αποτελεσματικά για να περιορίσει την κοινωτική χρηματοδότηση για να προωθηθεί το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ενετφέλτ για το Renew. Ναι, συγγνώμη, δεν σας είχα δει. Ήσασταν πρώτοι. Α, ε, δεν πειράζει, εντάξει. Ήδη έχω προαχθεί από την Άλντε στην ε, ομάδα Renew και έχω και χρόνο Ευχαριστώ πάρα πολύ την Επιτροπή για την ε, παρουσίαση και τη σύνταξη της ε, ετήσιας έκθεσης. Με χαρά άκουσα ότι λέτε ότι βελτιώθηκε χάρη στην ενθάρρυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Α, εντάξει, το λέτε ευγενικά. Εμείς πάντα ασκούσαμε κριτική και θεωρούσα ότι είναι ένα βασικό μέσο για να δημιουργηθεί μια κουλτούρα κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, κοιτώντας και την έκθεση που μόλις έχουμε λάβει, θεωρώ ότι η κριτική που εξέφρασα τα προηγούμενα χρόνια εξακολουθεί να ισχύει. Ότι δηλαδή η μέθοδος που χρησιμοποιείται δεν είναι αρκετά καλή και εξακολουθεί να βασίζεται πολύ στα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη τα ίδια. Οπότε, βασικά, Ε, σας δίνουν τα στοιχεία για μια έκθεση που υποτίθεται ότι θα κοιτάει με επικριτική σκοπιά τα κρατημέλη. Τώρα λέτε στην Πολωνία υπάρχουν κάποιες ανησυχίες. Είναι και πολύ ευγενικό. Θυμάμαι ότι είχαμε κάποιες ανησυχίες για την ε, Ουγγρική δικαιοσύνη και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Ε, στην έκθεση όμως ήταν μια χαρά όλα. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο κενό μεταξύ της εκθεσής σας και της πραγματικότητας, όπως το βλέπουμε όχι μόνο εμείς, αλλά οι πολίτες. Δηλαδή, αν μιλάτε για την ανάγκη εμπιστοσύνη στο σύστημα, χρειάζεται μία έκθεση η οποία θα δείχνει την πραγματική κατάσταση στα κράτη-μέλη σήμερα. Οπότε, σας παρακαλώ, για τον επόμενο πίνακα, ε, φύγετε από αυτή τη μέθοδο, μην βασίζεστε στα κράτη-μέλη, χρησιμοποιήστε κάποια άλλη πηγή ιδιαίτερος καθώς δεν είναι ε, κάτι το ετήσιο ένα κομμάτι χαρτί αλλά χρησιμοποιείται από τον μηχανισμό της ε, ρεσιμότητας. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Η έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για να κρίνουμε τα κράτη-μέλη και το εάν συμμορφώνονται και το εάν θα πάρουν τα κονδύλια. Είναι άχρηστη. Λοιπόν, εκτιμώ όλη τη δουλειά που έχει γίνει εδώ και τις καλές προθέσεις, αλλά δεν αρκεί. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι δική σας επιλογή. Είναι μια πολιτική επιλογή της Κομισιόν ενσώματι γιατί δεν θέλουν να τσαντήσουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Έτσι δεν είναι. Και γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν βλέπουμε πώς το Συμβούλιο έχει ορίσει όχι μόνο την πρόεδρο της Κομισιόν αλλά και τους άλλους επιτρόπους και το πώς εμπλέκονται πολύ ενεργά στην επιλογή χαρτοφυλακίων. Αυτό είναι ο λόγος. Είναι κρίμα ότι πρέπει να το συζητήσουμε τώρα με ελάχιστους βουλευτές παρόντες. Θα ήθελα να ζητήσω από τον πρόεδρο να το ξαναφέρει και να συζητήσουμε όχι μόνο τα αποτελέσματα αλλά και την μεθοδολογία και να ζητήσουμε από την Κομισιόν να αλλάξει μεθοδολογία για το επόμενο έτος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν έχει κάποιο ώρας να πει κάτι. Κανείς. Όχι. Παρακαλώ. Ναι, θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτό το οποίο είπε η κυρία Ινετφέλντ. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν επαγγελματία ε, ελεγκτής ε, τη φλαμανδική ε, διοικηση. μια διοίκηση ικανή και επαγγελματική. Και μα λέει τώρα ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη διοίκηση των κρατών μελών η κυρία Ινετφέλντ. Αυτό είναι απλά μια δυσπιστία η οποία πραγματικά είναι σκοφαντία κατά των εθνικών δημοκρατίων και εθνικών διοικήσεων οι οποίε λειτουργούν. Ναι, κυρία Ινετφέλντ. Εντάξει, καλή εμπιστοσύνη, αλλά ο έλεγχος είναι καλύτερος. Θεωρώ ότι η δημοκρατία πρέπει να έχει δικλείδες ασφαλείας. Αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας και όχι η τυφλή εμπιστοσύνη σε οποιαδήποτε εθνική διοίκηση. Λοιπόν, στην Κομισιόν τώρα, αν δεν θέλει κάποιο άλλο κάτι άλλο, κύριε Μπέλ, για να κάνετε τις τελευταίες σας πατήσεις. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως καλό είναι να θυμίσουμε πάλι τι είναι αυτός ο πίνακας ε, επιδόσεων και τι δεν είναι. Παρέχει μια συγκριτική εικόνα για τα εθνικά δικαστικά συστήματα και προσπαθεί να βοηθήσει την Ένωση και τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δικαστικών μεταρρυθμίσεων, παρέχοντας στοιχεία για την αξιολόγηση της ε, ποιότητας ανεξάρτησίας και της αποδοτικότητας, ε, αποτελεσματικότητας της ε, δικαιοσύνης, καθιστά ευκολότερη ευκολότερο τον εντοπισμό μειονεκτημάτων, την εξέβρεση λύσεων και να την παρακολούθηση των προκλήσεων και της προόδου που έχει γίνει. Είναι μια πρόσκληση στα κράτη-μέλη, στους ενδιαφερόμενους, εμπλεκόμενους φορείς να σημειώσουν τα αποτελέσματα και να ε, προβληματιστούν για στο, τους λόγους στους οποίους οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα, αλλά και στο να εντοπίσουν καλές πρακτικές, να στηρίξουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, των καλύτερων πρακτικών ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, τα δικαστικά του συστήματα. Εάν ε, ο πίνακας βαθμολογίας ε, δείχνει χαμηλές επιδόσεις, ε, εκεί θα πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτό, αυτή η βαθμολογία, να αναλυθούν βαθύτερα τα αίτια Και αυτό ε, και στη διαδικασία του εξαμήνου με το, για διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, το δικαστικό τομέα και εις βάθος ανάλυση της κατάστασης του δικαστικού συστήματος ε, που ε, εξετάζεται. Και ε, και λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες του δικαστικού συστήματος στο πλαίσιο του, ε, που ισχύει στο κάθε κράτος μέλος και αυτό μπορεί να οδηγήσει την Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμένου να προτείνει στο, στο Συμβούλιο να υιοθετήσει ειδικέ συστάσεις για ένα χώρα σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα. Έχουν υιοθετηθεί ε, ειδικέ ε, συστάσεις αναχώρα για 7 κράτη και προετοιμάζονται και άλλες. Υπήρξε και μια ερώτηση για το κατά πόσο αυτή η Επιτροπή το και το Κοινοβούλιο έχουν στηρίξει την εργασία του πίνακα του βαθμολογίου. Εγώ ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωκοινοβούλιο στις 29 Μαΐου πέρυσι ε, για το βαθμολόγιο του 2017 Κατά τη γνώμη μου αυτό το ψήφισμα ε, υποστηρίζει σαφώς, βεβαίως περιλαμβάνονται συστάσεις για βελτιώσεις για τις οποίες είμαστε πάντοτε ανοιχτοί. Πρόκειται για ένα εξελισσόμενο εργαλείο και προσπαθούμε πάντα να το βελτιώνουμε. Αυτό είναι σαφές. Αλλά αυτό το κάνουμε με την επικοδομητική στήριξη του Κοινοβουλίου. Έγινε μια ερώτηση για το ξέπλυμα χρήματος και για τις μακροσκελείς διαδικασίες σε αυτό το τομέα. Πρόκειται για πρώτη φορά που το βαθμολόγιο μπαίνει σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Για Έχουμε το, το σχέδιο 19 του πίνακα του βαθμολογίου που εξηγεί ακριβώς τι μετράτε εδώ. Πρόκειται για το μάκρος των δικαστικών υποθέσεων ε, στο πρωτοδικείο που βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ε, στα κράτη-μέλη και πάλι πρόκειται για μια, ένα θέμα σημαντικό ε, και περίπλοκο. Πάντως καλεί τα κράτη-μέλη να σκεφτούν το, τις διαδικασίες που ακολουθούν στο δικαστικό του σύστημα όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος ε, και βεβαίως θα τονίσουμε και πάλι αυτό το θέμα στις επόμενες εκδοχές, ε, ε, εκδόσεις μάλλον του βαθμολογίου. Τώρα για την ποιότητα της κρίσης και των αποφάσεων αυτό αυτή η πρόκληση είναι πολύ δύσκολη. Πώς δηλαδή δουλεύουμε με στοιχεία δεδομένα που εν γέννη ε, θεωρείται πως έχουν θετικό αντίκτυπο για τη, στην ποιότητα της, των αποφάσεων. Δηλαδή το πόσο που ε, έχει στον προπολογισμό του κάθε κράτος μέλος για το δικαστικό σύστημα, ε, αυτό μετράται, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο στην ποιότητα της δικαιοσύνης ε, και είναι κάτι συγκρίσιμο. Και αυτό το βλέπουμε μέσα στο βαθμολόγιο ως βάση για περαιτέρω προβληματισμό και συζήτηση για να βελτιώσουμε το δικαστικό σύστημα του κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπέλ, ευχαριστούμε για την παρουσίαση, ευχαριστούμε για την εργασία σας, για το ωραίο αυτό έγγραφο που είναι χρήσιμο εργαλείο και που στόχο έχει να ανταποκριθεί στο αίτημα της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ φρόντισε να υπάρξει ένα τέτοιο μέσο διαθέσιμο στα μέλη ε, για όσους ε, επιθυμούν να έχουν ε, συγκριτική νομική ανάλυση, να γνωρίζουν δηλαδή καλύτερα πώς λειτουργεί και ποιο είναι το δικαστικό τοπίο στη μελη ε, Και λοιπόν, τώρα προχωράμε. Χωρίς ε, άλλη καθυστέρηση, έχουμε ακόμα ένα σημείο να εξετάσουμε. Είναι μια ε, παρουσίαση, είναι το σημείο 12. Κοινοβουλευτική εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για να πάψει η κράτηση παιδιών μεταναστών. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Λα Φρεντές, που είναι Γενικός εισηγητής για την κοινοβουλευτική εκστρατεία αυτή και μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό για τον τερματισμό της κράτησης παιδιών μεταναστών και την προώθηση εναλλακτικών λύσεων είναι αυτό στην καρδιά της εργασίας μας. Το Ευρωκοινοβούλιο τον Μάιο του 2018 με ψήφισμά του για την προστασία των παιδιών μεταναστών δήλωσε την άποψη ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να προβεί σε διαδικασία κατά παράβαση ενάντια κρατών μελών για την συστημική κράτηση παιδιών μεταναστών και των οικογενειών τους, ώστε να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Γι' αυτό καλέσαμε εδώ τον κύριο Φριντές, που είναι ο Γενικός Εισηγητής για αυτή την κοινοβουλευτική εκστρατεία που γίνεται από την Κοινοβουλευτική Σύνοδο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μεταξύ σα, Μεγάλη μου τιμή κυρίω, διότι είμαι Ελβετός και δεν είναι συχνό φαινόμενο ένα ελβετό να έρχεται και να μην παίρνει το λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιο είναι το πλαίσιο λοιπόν αυτή τη εκστρατεία, Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια περίπου στο Συμβούλιο τη Ευρώπη σε ένα όλο ιδιαίτερο πλαίσιο αυτό του πολέμου της Συρίας, αυτό των εκατομμυρίων ανθρώπων που βρίσκονταν στους δρόμους με το δράμα που όλοι γνωρίζουμε και ανάμεσα στους μετανάστες όλους αυτούς υπήρχαν παιδιά, παιδιά πάρα πολλά, μη συνοδευόμενα, πολλά έχουν εξαφανιστεί και φανταζόμαστε εύκολα τι έχουν υποφέρει και πόσες δυσκολίες έχουν αντιμετωπίσει αυτοί οι άνθρωποι. Τον Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε η εκστρατεία στο Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από ένα ψήφισμα που είχε το εξή στόχο. Έλεγε λοιπόν πως δεν είναι ποτέ το συμφέρον ενός παιδιού να τοποθετείται να βρίσκεται υποκράτηση λόγω του καθεστώτος του ή του καθεστώτος των γονιών του. Πρόκειται για κράτηση ενώ δεν υπάρχει έγκλημα ή αδίκημα. Είναι μόνο ένα πρόβλημα που σχετίζεται με τη μετανάστευση και με τα ε, έγγραφα, δηλαδή μια διοικητική κατάσταση κατάσταση. Δεν μπορεί να κρατώνται παιδιά για λόγους μετανάστευσης. Θα έπρεπε καταρχάς τα παιδιά να αντιμετωπίζονται σαν παιδιά. Τα παιδιά είναι για να παίζουν, για να μαθαίνουν. Ε, ε, πρέπει δηλαδή οι ανήλικοι να αντιμετωπίζονται ως ανήλικοι, όποιο και να είναι το καθεστώς τους. Ε, ε, ε, θα έπρεπε να θελήσαμε να προσαρμόσουμε τη διαδικασία αξιολόγηση του ηλικία όσον αφορά τα παιδιά μεταναστών. Και κυρίω θέλαμε για τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου τη Ευρώπη να υιοθετήσουν εναλλακτικέ λύσει στην κράτηση που να ανταποκρίνονται στο ανώτατο συμφέρον του παιδιού, δηλαδή σε ένα μη ε, σοφρονιστικό περιβάλλον τα παιδιά μεταναστών είτε είναι συνοδευόμενα είτε όχι είναι συχνά η πιο ευάλωτη ομάδα ανάμεσα από όλους τους μετανάστες και η κατάστασή τους μπορεί πολύ γρήγορα να γίνει πολύ δραματική. Ένα ουσιαστικό στοιχείο αυτής της εξαρτίας ήταν η προβολή όλων των ε, θεμάτων υγείας που μπορεί να συνδέεται ε, με, αυτά. Εγώ είμαι γιατρός, είμαι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε αυτή την κατάσταση και θεωρούμε πως η κράτηση μπορεί να έχει πολύ σημαντικές συνέπειες στην υγεία και την ανάπτυξη ενός παιδιού. Το γεγονός ότι είναι κλεισμένο ε, μέσα κάπου δεν μπορεί να το επηρεάσει, κυρίως όταν δεν καταλαβαίνει το γιατί και το πώς. Μπορεί να οδηγηθεί σε απόπειρες αυτοακροτηριασμού αλλά και ε, αυτοκτονίας. Ένα παιδί με χαρακές στα χέρια του ε, είδα σε ένα καταβλισμό προσφύγων στην Ουγγαρία όπου κρατοκτήτω το για πολλούς μήνες. Μπορεί να έχει προβλήματα ύπνου, προβλήματα ανάπτυξης ε, κοινωνικοποίησης ψυχολογικά, ανάπτυξη εξι προβλήματος ε, ε, ε, ε, ψυχολογικού. Δεν είναι ποτέ ανώδυνο. Μπορεί να έχουν ε, ακράτεια ούρων, μπορεί ε, οτιδήποτε να του συμβεί. Επίση δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Συχνά χάνουν το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση ή το δικαίωμα για κάποιο προστάτη, κάποιο που βρίσκεται εκεί για να του βοηθήσει. Το δικαίωμα στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Τα παιδιά αυτά μπορεί να παραμεληθούν και να υποστούν κατάχρηση ενώ ήδη έχουν εκτεθεί σε βία. Ε, φρικτή στη διάρκεια του ταξιδιού του. Στην Ελλάδα, σε ένα σπίτι όπου ε, υποδέχονταν παιδιά σε φανταστικές συνθήκες, είδα ένα νεαρό κορίτσι 13 ε, χρονών που ήταν έγκυος μετά από βιασμό. Ε, ε, στόχος ήταν λοιπόν να ευαισθητοποιήσουμε τα χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης σε αυτά τα προβλήματα και κυρίως να ευαισθητοποιήσουμε τους βουλευτές για αυτή την κατάσταση ώστε να μπορέσουν να ενημερώσουν στις χώρες τους για να εξελιχθούν και οι σχετικές νομοθεσίες. Κάναμε λοιπόν έρευνες όσον αφορά την πρακτική, κυρίως για τις χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει σχετικέ εργασίες που σίγουρα θα τι γνωρίζετε και εκπονήσαμε έναν οδηγό για να βοηθήσουμε τους βουλευτές αλλά και άλλους να μπορούν να κάνουν επισκέψεις σε ιδανικέ συνθήκε, γιατί υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που πρέπει κανεί να σκεφτεί όταν πάει σε μια φυλακή ή σε κάποιο κέντρο κράτησης. Σε αυτή την εκστατεία επισκεφθήκαμε ένα σωρό δομές που ε, στέγαζαν παιδιά. Ας πούμε, ε, επισκεφθήκαμε ένα καταβλισμό ε, προσφύγων στο Ζάταρι στην Ιορδανία. Ήταν ιδιαίτερα η κατάσταση γιατί ήταν μόνο Σύριοι στα σύνορα με την Συρία. Ήταν σχετικά καλή κατάσταση. Είδαμε ένα, ένα καταβλισμό προσφύγων στην Αυστρία, στην Ουγγαρία στο Ρέσκε, όπου η κατάσταση ήταν πολύ πιο περίπλοκη και επισκεφθήκαμε κυρίως για να δείξουμε στους βουλευτές τι μπορούμε να κάνουμε ε, εγκαταστάσεις ε, στα κάτι μέλη που ισχύαν πολύ καλές πρακτικές όσον αφορά ε, τα παιδιά τα, μη συνοδευόμενα. Δεν έχουμε ε, μια ομοιόμορφη προσέγγιση, αλλά μια προσέγγιση ανά περίπτωση όπου κάθε παιδί έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Το κάναμε αυτό στην Ελλάδα, στην Ελβετία, στην Κύπρο και εδώ θα ήθελα να σας προτείνω να δούμε ένα βίντεο ε, ε, ενός κέντρου στην Ελβετία που είναι ένα κέντρο αριστείας αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Φριντές. Σας ευχαριστούμε που κάνατε αυτή την εκστρατεία. Α, θα συνεχίσω μετά, θα έχω και άλλα να σας πω μετά το βίντεο. Μάλιστα, θα δούμε το βίντεο και μετά θα συνεχίσετε. Ωραία. I've been Μου είπαν ότι το βίντεο αυτό που δείχνει την εξατία θα είναι μόνο στα αγγλικά. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους που δεν θα μπορέσουν να έχουν μετάφραση. Είναι στα αγγλικά το βίντεο λοιπόν.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 I'm working like let me say four years now. All these four years I was experiencing that some of them they even go far chill to Bern to find uh, clubs where they play basketball, volleyball. من میخوام سپورت پولونی را کنم به خاطرش که در افغانستان اونمو کلتور ماست دیگه دیگه اونمو را بسیار دوست دارم دیگه غیر از او سپورت های دیگه را انجام دادیم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 Ορίστε, το επισκέφθηκα αυτό το κέντρο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση το πιο μικρό παιδί ήταν 6 ετών. Ένα νεαρό Αφγανό που είχε έρθει με ένα αδέλφι 10 ετών. Όταν βλέπουμε αυτέ τι καταστάσει, ξέρουμε πω αυτά τα παιδιά θα μείνουν στη χώρα μα. Άρα μα συμφέρει να αγωνιστούμε και να του εξασφαλίσουμε ένα μέλλον, να μάθουν τη γλώσσα, να μπορέσουν να ενσωματωθούν, πάνε στο σχολείο του χωριού μαζί με τα παιδιά του χωριού και από τη στιγμή που κάπως μιλάνε τα γερμανικά και προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε για κάθε παιδί ε, ε, ε, πρόγραμμα στα μέτρα του. Στην Ελλάδα, όπου η κατάσταση οικονομική είναι πιο δύσκολη και ορισμένα παιδιά θέλουν να φύγουν αλλού, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να προσπαθήσουμε να του βρούμε σε μια άλλη χώρα κάποιον από την οικογένειά του για να κάνουμε οικογενειακή επανένωση. Δηλαδή, για τον καθένα προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα στα μέτρα του. Τώρα, να σα πω ότι αν είστε ενήλικο, δεν, σας μεταχειρι... δεν μπορούν να σα μεταχειρίζονται σαν να είστε ενήλικο. Ο νόμο αλλάζει τελείω. Το παιδί προστατεύεται ενώ ο ενήλικας πολύ λιγότερο και μάλιστα σε ορισμένες χώρες η αξιολόγηση της ηλικία γίνεται κάπως αυθαίρετα. Ε, λέει ότι υπάρχει αυτό που λέει το παιδί, αλλά δεν υπάρχουν πάντοτε έγγραφα. Είναι παιδιά που έρχονται ας πούμε από, από, χώρες που επικρατούν συνθήκες πολέμου, δεν έχουν τα χαρτιά που πρέπει μαζί τους. Λένε ότι έχουν κάποια ηλικία, αλλά συχνά αυτό είναι αμφισβητήσιμο. Πώς κάνουμε λοιπόν, υπάρχουν μέθοδοι τελείως άχρηστες. Εγώ σας μιλώ σαν γιατρός, ας πούμε γίνονται ε, ακτινογραφίες. Ακτινογραφία της ε, παλάμης του χεριού και με βάση ορισμένα κόκαλα μπορούμε θεωρητικώς να δώσουμε μια ηλικία αλλά πάνω κάτω μπορούμε να πέσουμε έξω ε, ε, τρία χρόνια πάνω τρία χρόνια κάτω δηλαδή άμα πούμε ότι είναι 17 ετών μπορεί κάποιος να είναι στην ουσία από τα 14 μέχρι τα 20 στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ μεγάλη ακρίβεια. και αυτό μπορεί να στιγματίσει τα παιδιά για το Συμβούλιο της Ευρώπης εμείς κάναμε ένα ψήφισμα που λέει ότι σε κάθε περίπτωση η αμφιβολία όσον αφορά το αν είναι ανήλικο το παιδί, όχι, θα πρέπει να ωφελήσει, το, να είναι υπέρ του παιδιού. Εμείς λοιπόν εξακολουθούμε ε, να κάνουμε αυτές ε, τις εκστρατείες ε, για να τελειώσει η βία, να σταματήσει η βία και η εκμετάλλευση επί των παιδιών, μετα, παιδιών μεταναστών. Η σεξουαλική βία είναι κάτι το φρικτό και ασκείται συχνά στα παιδιά. Ε, θέλουμε να φτιάξουμε ένα μέσο που να προστατεύει το κάθε παιδί, το μη συνοδευόμενο παιδί μετανάστη, να μπορεί να έχει έναν προστάτη που θα υπερασπίζει τα συμφέροντά του. Τέλο, μιλάμε εδώ για παιδιά τα οποία δεν έχουν ε, διαπράξει κανένα αδίκημα ε, ούτε έγκλημα, η ευημερία του παιδιού είναι αυτό που θα πρέπει να έχει την πρώτη καθεδρία, ε, να, προ, να προωθηθούν μέτρα εναλλακτικά της κράτησης. Αν θέλετε μπορώ να σας πω κάποια περισσότερα πράγματα. Η κράτηση του παιδιού θα πρέπει να είναι κατεξαίρεση, να είναι κατά αναλογία και όσο γίνεται πιο σύντομη διάρκεια. Και κυρίως πρέπει να σκεφτούμε το μέλλον αυτών των παιδιών. Είμαι ευτυχής που μιλάω εδώ σε μια νέα στη νέα θητεία και θα ήθελα αυτό το θέμα να είναι προτεραιότητα για σας. Πρέπει να γίνει λοιπόν ε, αναπερίπτωση προσέγγιση και όχι μια ομοιόμορφη για όλα τα παιδιά. Να σας διαβάσω ένα κείμενο της Επιτροπής σας του 2017 που δίνει τη σύνοψη των όσων πρέπει να γίνονται. Αναγνώριση και αγρήγορη προστασία από την άφηξη μόλις. Προστασ... Ε, δομές υποδοχής κατάλληλες ε, με κέντρο υγείας και εκπαίδευσης Επίση, διοικητικέ διαδικασίες και αν πρέπει να περάσουν από κράτηση, δεν είναι πιο σύντομη γίνεται. Προστασία γρήγορη και αποτελεσματική. Αξιόπιστη και σωστή διαδικασία αξιολόγησης της ηλικία. Μέτρα πρώιμης ε, ένταξης. Ένα θέμα με ανησύχησε λίγο στις πληροφορίες που μου έδωσαν όσον αφορά την οδηγία της επιστροφής επί της οποίας εργάζεστε και φαίνεται πως στην αναθεώρηση της οδηγίας πάντοτε υπάρχει αυτή η ιδέα ότι θα υπάρχει δυνατότητα να κρατείτε ένα παιδί μέχρι και για τρεις μήνες. Το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, κυρίε και κύριοι, είναι θεμελιώδε, ακόμα περισσότερο για τα παιδιά. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Φρυδέ, για την εκστρατεία σα και ευχαριστώ που επιστήνετε την προσοχή μα σε αυτό το τόσο της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για αυτό το θέμα που είναι τόσο ευαίσθητο εμείς το συζητάμε και στα ψηφίσματά μας ε, μετά από την κρίση την μεταναστευτική. Είναι λοιπόν η προστασία των ε, ανήλικων στην καρδιά της Επιτροπής Λίγη. Τώρα έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση και χτες ε, ε, χρειάστηκε να, ευχαριστήσω θερμά τους διερμηνείς για την παράταση που μας έδωσαν για κάποια παραπάνω λεπτά, γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο μας το χτες. Ε, σήμερα ίσως και να χρειαστεί πάλι να ζητήσω λίγα περισσότερα λεπτά, γιατί μόνο 8 λεπτά μας έχουν μείνει. Ε, παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι, ώστε να μην εξαντλήσουμε τους διερμηνείς μας όπως και εχθές. Α, μέχρι τις 12.30 έχουμε. Α, εγώ νόμιζα πως ήταν μέχρι τις 12. Α, τότε εντάξει. Έχουμε τράτο, ε, ώστε να μπορέσετε να μιλήσετε. Κινίτσι πρώτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Φρυδές για την εισήγηση αυτή που μας κάνατε για την ε, εξατία υπέρ της προστασίας των ανηλίκων. Εσείς ε, θίξατε ένα θέμα ευτυχώς που εμένα μου είναι ιδιαίτερα ε, αγαπητό η προστασία των ανηλίκων στην οποία έχω αφιερώσει πάρα πολύ μέρος της δουλειάς μου ως εισαγγελέο, πριν να έρθω στο Ευρωκοινοβούλιο και τώρα στην προηγούμενη θητεία ως ιδρύτρια και πρόεδρος του Intergroup για τα δικαιώματα των ανηλίκων που δούλεψε πολύ, πάρα πολύ για τα θεματικές που αφορούν την προστασία των ανηλίκων αλλά και συγκεκριμένα στην προηγούμενη θητεία δουλέψαμε για τους ανήλικους μετανάστες και αντιμετωπίσαμε όλες αυτές τις πτυχές που αναφέρατε και εσείς. Ο Πρόεδρος Λόπες Αγγιγιάρα ανέφερε επίσης το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την προστασία των ανηλίκων του Μαρτίου 2018. Είναι αλήθεια η Επιτροπή μας όπως και το Intergroup εκεί συνέβαλαν όλος ιδιαιτέρως. Το θέμα της κράτησης των παιδιών των ανηλίκων μόνο λόγω του καθεστώτος τους ε, ως μεταναστών έχει συζητηθεί και στο φόρουμ για τη δικαιώματα των ανηλίκων που συγκάλεσε η Επίτροπος Γιούροβα και πριν από δύο ε, ε, χρόνια. Επιπλέον εγώ είμαι Ιταλίδα, είμαι και από τη Σικελία, οπότε καταλαβαίνετε χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε επιτόπου το θέμα της μετανάστευσης και εγκρίναμε και άρχισε να ισχύει μια, ένα ειδικό νόμο όσον αφορά τα μέτρα υποδοχή και στήριξη των παιδιών μεταναστών που φτάνουν ε, στην επικράτειά μα. Η καταδίκη ε, κατά τη κράτηση των παιδιών μεταναστών είναι σταθερή. Εγώ, επειδή έχω δουλέψει και ω εισαγγελέα σε αυτό το τομέα, ξέρω ποιε είναι οι συνέπειε τη κράτηση για τα παιδιά, ακόμα και αυτά που έχουν διαπράξει αδικήματα. Και γι' αυτό και πάντοτε Τότε σκεφτόμαστε εναλλακτικέ λύσει. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι απαράδεκτη λοιπόν η κράτηση ανηλίκων. Ε, καλό θα ήταν, καλύτερο θα ήταν να σα πω ότι έχουμε κάνει στη χώρα μου και στη χώρα εδώ ε, και εδώ εντός του Ευρωκοινοβουλίου καλό είναι να υιοθετηθούν ειδικά μέτρα υποδοχή και στηρίξή των ανηλίκων. Εσεί αναφέρθηκατε ήδη σε κάποια, Όπω είπατε πρώτα απ' όλα σωστή αναγνώριση και άρα εντοπισμό τη ηλικία του παιδιού ώστε να παρέχουμε την προστασία που αντιστοιχεί σε αυτή την ηλικία. Δηλαδή, ορισμό κάποιου προστάτη, εντοπισμό ανάμεσα στου ανήλικου που φτάνουν των όσων ας πούμε, έχουν πέσει θύματα τη εμπορίου, καταχρήσεων, βία, για να μπορέσουμε να δώσουμε, να προσφέρουμε το είδο τη υποδοχή και το είδο τη ε, αγωγή, θεραπεία ε, που αντιστοιχεί σε αυτέ τι δραματικέ καταστάσει που ίσω έχουν ζήσει. Και μετά μια ολόκληρη σειρά που εγγυώνται την κατάλληλη υποδοχή, τη θεραπεία, τη στήριξη και την κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών. Είδαμε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο που ακριβώς δείχνει πώς θα πρέπει να είναι αυτό το είδος στήριξης προς τα παιδιά μετανάστες. Ο χρόνος μας δεν είναι πολύ, οπότε υποχρεώμαι να κλείσω. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο με συναρπάζει και θέλω να ρωτήσω για να μπορέσουμε όντως να στηρίξουμε καλύτερα αυτά τα παιδιά. Κατά τη γνώμη σας, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια συνεργασία μπορούμε να κάνουμε μεταξύ ε, του Ευρωκοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ακριβώς ώστε να επιτύχουμε αυτό το στόχο, να ξεπεράσουμε την κράτηση και να δώσουμε πιο κατάλληλη στήριξη στα παιδιά μετανάστες. Ε, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησε, αλλά είναι ε, πολύ συναρπαστικό το θέμα. Μάλιστα, παρακαλώ έχετε τον νου στο χρόνο. Κυρία Ιντεβέλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς και εσάς κύριε Φρίντες, για την παρουσίαση του θέματος. Να κάνετε το ίδιο και στο Συμβούλιο. Αυτό θα σας συστήσω, διότι το θέμα της κράτησης παιδιών είναι από τα βασικά ε, ζητήματα που δεν επιτρέπουν να καταλήξουν σε ε, τελική συμφωνία. Γιατί οι χώρες μέλη φαίνεται να έχουν ένα είδος ε, Μανία να κρατούν ανθρώπους, μεταξύ αυτών και παιδιά. Και ναι, μεν επικρίνουμε τις φρικτές συνθήκες που βλέπουμε στις Ηνωμένε Πολιτείε, λησμονούμε ότι εδώ στην Ευρώπη και τα παιδιά κρατούνται και όχι μόνο οι ασυνόδευτοι ενήλικοι, αλλά και συνοδευόμενοι ενήλικοι. Και υπάρχει ένα πραγματικό δίλημα, δηλαδή, όταν βάζει κανείς τους γονείς σε κράτηση θα βάλει και τα παιδιά μαζί με τους γονείς ή θα χωρίσει τις οικογένειες, το οποίο επίσης είναι τραυματικό για τα παιδιά, για όλους δηλαδή. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είναι τόσο ε, αιμονικοί να κρατούν τον κόσμο, να τους βάζουν σε κράτηση δηλαδή, εκτός αν δεν υπάρχει άλλο μέσον. Γιατί βλέπουμε τις εθνικές κυβερνήσεις να επιμένουν σε κρατήσεις και κρατούν και ε, τους πάντε με τα παιδιά τους και καμιά φορά μάλιστα χωρί δικαστική παρέμβαση. Πρόκειται για διοικητικέ διαδικασίες, ε, Διοικητικέ ε, διαδικασίες για την κράτηση. Εγώ ήμουν μάλιστα εισηγήτρια για την σχετική οδηγία όπου μπορέσαμε υπό βουλγαρική προεδρία να διαπραγματευτούμε και τελικώ να καταλήξουμε σε μια λίγο πολύ αποδεκτή λύση. Είπαμε δηλαδή ότι κάθε φορά που υπάρχει απόφαση να κρατηθεί ένα παιδί θα πρέπει να επαληθεύεται από ένα δικαστή ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Και αυτό ακόμη που είναι βεβαίω και νομοθεσία των ΗΠΑ αμφισβητείται από τις εθνικές αρχές. Κάτι άλλο που προτείνουμε είναι ότι κάθε παιδί άμα τη αφήξει του να του ορίζεται ένας ε, πρόσωπος, νομικός εκπρόσωπος όχι μόνο και δαιμόνας, αλλά να, είμαστε, να είναι δηλαδή έτσι βέβαιο ότι κάποιος φροντίζει τα νόμιμα δικαιώματα του παιδιού. Και όπως είπε και προλαλή σα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κατ' επανάληψη ψηφίσει και με μεγάλη μάλιστα πλειοψηφία από αριστερά μέχρι δεξιά μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για να πούν ότι θα πρέπει να απαγορευτεί η κράτηση παιδιών. Απόλυτη απαγόρευση. Δηλαδή, ναι, μην έχουμε κάνει κάποιο δρόμο ε, για να ε, ε, μπορέσουμε να συνοηθούμε με το Συμβούλιο, αυτό σημαίνει μεγάλη παραχώρηση εκ μέρου μα. Δεν μπορούν οι χώρε μέλη να έχουν απεριοριστέ δυνατότητε να θέτουν τα παιδιά σε κράτηση. Γιατί έτσι κάνουμε ό,τι κάνει και η κυβέρνηση Τραμπ. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για όλα. Κυρία Στρίκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Φρίντες. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που βλέπω ένα πρώην συνάδελφό μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ ήμουν μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης από τον προηγούμενο μήνα. Είμαι μάλλον. Στο δεύτερο που έρχεται τώρα εδώ στην Επιτροπή ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών, εγώ είχα μάλιστα έρθει τότε το 2012 για τους θανάτους που σημειώνονται στη Μεσόγειο και τώρα έρχεται, έρχεστε εσείς για την κράτηση παιδιών. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ε, τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών συνελεύσεων. Είμαι και ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την παρουσίαση της εκστρατείας, διότι πράγματι νομίζω ότι απηχεί μια κοινή, αίσθηση παγκοσμίω ότι η κράτηση παιδιών είναι, αποβαίνει πάντοτε εις βάρος τους και ποτέ δεν είναι προς το συμφέρον τους. Μπορώ ίσως να σας εξηγήσω και μερικές από τις εμπειρίες που είχα συλλέξει από την κοινοβουλευτική συνέλευση, διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης τελικώς, το Υπουργικό Συμβούλιο δηλαδή, αποφάσισε να συντάξει στις στάσεις για τις κρατήσεις, ίδιες όπως και για τις φυλακίσεις, αλλά μόνο για, αυτές ισχύουν όμω μόνο για ε, ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί Ο μόνο λόγο για τον οποίο κρατούνται ε, μετανάστες είναι για να μην εξαφανιστούν. Ε, χρειάζονται λοιπόν άλλοι κανόνε. Είχα συμμετάσχει στι διαπραγματεύσει αυτέ και είχαμε κάνει σημαντική πρόοδο και μόλι στο τέλο τη διαδικασία αυτή παρενέβη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι διαπραγματεύσει εξ ονόματο, όπω είπε, των χωρών μελών και ζήτησε σημαντική αποδυνάμωση των προδιαγραφών. Είπε ότι θέλει να καταργήσει όλες τις διαδικαστικές εγγύησεις, να καταργήσει την ε, αρχή ότι δεν θα κρατούνται παιδιά, ότι δεν θα κρατούνται έγκυες γυναίκες και βέβαια εν τέλει, διότι η πλειοψηφία των χωρών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η πλειοψηφία, είναι οι χώρες μέλη της Ένωσης. Τελικώς αναστάλησαν οι ε, διαπραγματεύσεις αυτές και φτάσαμε εκεί που έχουμε φτάσει. Και αυτό νομίζω είναι πραγματικά ένα σκάνδαλο ότι συνέβη αυτό. Για διαφόρους λόγους. Ένας είναι ότι εγώ θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεπερνούσε μάλιστα το Συμβούλιο της Ευρώπης. Διότι το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να προτείνει ελάχιστες ε, προδιαγραφέ για τι 47 χώρε μέλη του ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ψηφίσει πραγματική νομοθεσία. Είναι λοιπόν απίστευτο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα καταφέρνει και αποδυναμώνει τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και λυπούμε πολύ, διότι και οι χώρε μέλη εξαρτώνται από, αυτές, από αυτούς τους κανόνες. Και σωστό είναι να επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε και οι υπόλοιπε χώρες που δεν είναι μέλη της, να αυξήσουν τα πρότυπά τους. Υπάρχει και ένα θέμα δημοκρατική νομιμοποίηση. Εγώ εκεί εκπροσωπούσα το PACE. Είμαι βεβαία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην παρέμβασή τη εκείνη. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για μα. Τώρα, να τελειώνω σιγά σιγά. Υποστηρίζω την εκστρατεία σα. Ελπίζω ότι θα τα λάβουμε υπόψη αυτά και στι τρέχουσε διαπραγματεύσει. Και η κυρία Ιντφέλτ μίλησε για το ψήφισμα που εγκρίναμε την προηγούμενη εβδομάδα και το οποίο λέει ότι η κράτηση παιδιών δεν είναι ποτέ προς το πραγματικό συμφέρον τους και ελπίζω αυτό να ενθαρρύνει την επίτευξη ενός πραγματικού αποτελέσματος για το Κοινοβούλιο και το ρόλο που θα παίξει στην οδηγία επιστροφών. Είχαμε πει αρχικώς μέχρι τις 12 και ναι, μεν δεχόμαστε ευχαρίστως την παράταση, αλλά εγώ έχω ε, συνάντηση στις 12 και 4 με τον ε, Υπουργό Δικαιοσύνη της Λιθουανίας. Ελπίζω να προλάβω. Θα χρειαστώ τη βοήθειά σας όμως, ο κύριος Μαγκίντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος και σας ευχαριστώ και σας αγαπητέ για την παρουσίασή σας. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού έχουμε φρικιαστικές σκηνές στα σύνορα με το Μεξικό. Βλέπουμε τις νοοτροπίες που σκληραίνουν και για τα παιδιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως είπατε και εσείς στις 13 Αυγούστου στο Ελβετικό ραδιόφωνο, σωστά μιλήσατε για το ψυχολογικό τραύμα των ασυνόδευτων παιδιών ε, που κρατούνται. Ε, ε, Μπορεί να μετρήσετε εσείς ποιον αντίκτυπο θα έχετε, αλλά μήπως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να τριπλασιάσει τους πόρους τους ε, και να αναλάβουν την ηθική ευθύνη να σταματήσει η κράτηση παιδιών στην Ήπειρό μας και να το πάμε και στις ΙΠΑ ε, γιατί πρόκειται για μια παράδεκτη πρακτική απέναντι στα παιδιά μετανάστες και μιλάμε εδώ πέρα για παιδιά. Δεν πρέπει να παραμελήσουμε και τους 19χρονους και 29χρονους που μόνο κίνδυνο έχουν γνωρίσει και δεν έχουν ακόμα οριμάσει και χρειάζονται και αυτή η στήριξη όπως τα παιδιά. Ε, άμα είναι να μεγαλώσει ο κατάλογος θα μπλέξω κι εγώ. Παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ναι, ναι. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα υπόθηκαν. Είναι σαφές ε, πως ε, μας ανησυχεί και προβληματίζει ιδιαίτερα το πρόβλημα και θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Φιντές για την ε, έκθεση που μας κάνατε και για το γεγονός ότι σήμερα το συζητάμε. Εγώ είχα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν να ρωτήσω αν υπάρχουν εκθέσεις για τις διάφορες χώρες, αναχώρα για το πώς αντιμετωπίζετε το θέμα και επίσης να δούμε πώς θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα καλά παραδείγματα, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα, και πώς μπορούμε να τα διαδώσουμε. Αυτά τα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρικμοντ, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Φιδές. Η ομάδα μας 100% ε, συμφωνεί με τις συστάσεις και την εξαρτία που κάνετε. Είναι μια ευκαιρία για να ευαισθητοποιήσουμε, αλλά πώς θα προχωρήσουμε πέρα από αυτό, γιατί διαπιστώνουμε τη, την υπεχρέωση κρατών όπως το Βέλγιο, η Γαλλία, το Υπουργείο Εξωτερικών μόλι αποφάσισε να ξανακλείσει ε, παιδιά στο κέντρο ε, Μπις, σε, σε, Μπις, ακριβώς έξω από το Ζάβεντε, με φρίκη οι συνθήκες εκεί, παρά τις εκθέσεις και παρά τις εξαρτίες ευαισθητοποίησης, ε, τα κράτη-μέλη είναι αυτά που κλείνουν παιδιά στις φυλακές. Πώς λοιπόν μπορούμε να, δώσουμε, να διαδώσουμε αυτή την εκστρατεία, υπάρχουν εκστρατείες. Στο Βέλγιο, ας πούμε, να, θα μπορούσε να λέει, δεν γίνεται γίνεται να ε, φυλακίσεις ένα παιδί. Ε, ε, μπορούμε να κάνουμε εξατίε και να μπορέσουμε να αγγίξουμε έτσι τις κυβερνήσεις και τα κάτι μέλη. Ευχαριστώ κυρία Κένκο. Ευχαριστώ. Το ερώτημά μου είναι πράγματι πάρα πολύ σύντομο. Λοιπόν, το ερώτημα μου είναι ακούμε όλα αυτά τα πράγματα για την ε, κατάσταση των ε, παιδιών ε, αλλά δεν ακούμε τίποτα για την ευθύνη των χωρών προέλευσης γιατί αυτό σημαίνει ότι κάποιος κάπου δεν έχει κάνει την δουλειά του. Λοιπόν, εμείς μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά βλέπουμε επί σειρά ετών τα ίδια προβλήματα όταν κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν τη δουλειά. Μιλάω για τους ηγέτες συγκεκριμένων χωρών που δεν προστατεύουν ε, τους ε, λαούς τους. Και δεύτερον, ε, βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια που είναι θύματα όχι μόνο σε αυτές τις ε, διαδικασίες αλλά και στις ε, χώρες προέλευσης και σε ευρωπαϊκό έδαφος που είναι ανήλικες και αναγκάζονται να γίνουν νύφες. Ε. Και τέλος, ε, πράγματι είναι πάρα πολύ σοβαρές οι συνθήκες και αυτό οφείλεται και στην έλλειψη μιας πραγματικά ευρωπαϊκής ε, μεταναστευτικής ε, πολιτικής. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. There... Κάποιος άλλος? Ναι, ναι, σύντομη ε, τότε παρακαλώ να είστε. Ναι. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν κάποιες φρικτές ανθρωπιστικές καταστάσεις, ειδικά οι ανθρώπους που έρχονται παρανόμως στην Ευρώπη. Για εγώ είμαι πατέρας δύο μικρών παιδιών και είχα δει το 2015 αυτές φρικτές εικόνες του Αϊλάν και μη είχε ρωτήσει τότε ο γιος μου «Ε, «Μα γιατί» είπε τον ε, άφησε ο πατέρας του. Πράγματι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από ε, καταπιεστικά καθστώτα και πράγματι θα έπρεπε επί της αρχής να μην κρατούνται ε, άνθρωποι, αλλά όταν με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ένας διάβλος ε, παράνομης ε, μετανάστευσης, βλέπουμε αυτό το οποίο έχουμε στο Βέλγιο, που αυξάνει ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που έρχονται στην Ευρώπη. Και μετά έχουμε το σύστημα της οικογενειακής επανένωσης, που δημιουργεί έτσι έναν διάβλο, όπως είπα. Οπότε, το ερώτημά μου τελικά είναι Ε, μήπως ε, έτσι με αυτόν τον τρόπο τελικά παρακινούμε ειδικά την ε, παράνομη μετανάστευση, ειδικά των αλήκων. Θα απαντήσω πρώτα στις ε, δύο τελευταίες παρεμβάσεις που τοποθετούνται σε διαφορετικό πλαίσιο. Ευθύνη των χωρών ε, προέλευσης. Ναι, αυτό είναι προφανές. Ωστόσο, η παγκόσμια πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν χώρες ε, σε εμπόλεμη κατάσταση, υπάρχουν δικτάτορες, δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε αυτό. Εμείς είμαστε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Αν ο Σύριος δικτάτορες ε, είχε φερθεί σωστά, ε, θα είχε ίσως λυθεί το πρόβλημα πιο εύκολα και δεν θα χρειαζόταν τώρα σε πόλεμα. Έπειτα υπάρχει κλιματική αλλαγή. Όλο και περισσότερος κόσμος θα μετακινείται. Μετά έχουμε ε, και δημογραφική ανάπτυξη. Ένα δις είναι στην Αφρική αυτή τη στιγμή, ενάμιση θα είναι το 2050 και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος μετακινείται για να βιβιώσει. Ε, ε, αυτό θα απαντήσω στον τελευταίο ομιλητή. Εξορισμού αυτή η μετανάστευση είναι πάντοτε παράνομη, γιατί προσπαθούν να σωθούν και κινούνται. Υπάρχει απειλές, πόλεμος, πείνα, ε, δικτάτορες προσπαθούν να φύγουν για να τα καταφέρουν. Η χώρα μου, η Ελβετία, το 19ο αιώνα είχε πάρα πολύ μετανάστευση, κυρίως στην Λατινική Αμερική, γιατί δεν υπήρχε δουλειά τότε στην Ελβετία είναι ανθρώπινο. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Όλοι όμως θα ε, ε, πρέπει να φροντίσουμε να συμπεριφέρονται ανθρώπινα. Ε, και σωστά. Και ένα παιδί είναι ένα ανθρώπινο όν που πρέπει να προστατευτεί γιατί υπάρχει το μέλλον του. Εάν το μεταχειριστεί άσχημα τον κόσμο που φτάνει στην χώρα σου, στην ουσία στρώνεις στο δρόμο για άλλα πράγματα, για κρεότητες, για τρομοκρατία. Ε, ε, πρέπει δηλαδή να τους δεχτούμε με το σωστό τρόπο. Κυρία Κινίτσι, η συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Ναι, είναι προφανέ. Όμω, ανάμεσα στι δύο κοινοβουλευτικέ συνελεύσει υπάρχουν μια μεγάλη διαφορά και ζητώ συγγνώμη για αυτό που θα πω για του συναδέλφου του Συμβουλίου τη Ευρώπη, όπου ήμουν ε, ε και εγώ μέλο. Είπα... Εμεί είμαστε κάπω μια λέσχη που αγωνίζεται για να προχωρήσουν προς τα πάνω τα ανθρώπινα δικαιώματα, η σεβασμό της δημοκρατίας στο κράτος δικαίου. Αλλά κάνουμε μόνο συστάσεις, ενώ εσείς ε, είστε μια κοινοβουλευτική συνέλευση που λαμβάνει αποφάσεις, φτιάχνει νόμους, ε, ε, κανόνες. Εσείς θα πρέπει να αποτελέσετε την κινητήριο δύναμη, τη μηχανή. Εμείς μπορούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να το ζητήσουν ε, γενικώς και να το εφαρμόσουν γενικώ και ορίστως. Εμείς πάμε στα... μέχρι και στην άκρη της Ασίας. Υπάρχουν χώρες που είναι πιο γρήγορες από τις άλλες, ναι. Αλλά πιστεύω πως ο δικός σας ρόλος είναι καθοριστικός. Κάποιο ρώτησε σε σχέση με το ποιες είναι οι σχέσεις, ε, οι εκθέσεις με συγχωρείτε, για τις διάφορες χώρες. Εδώ ε, το Συμβούλιο της Ευρώπη έχει φτιάξει μια έκθεση. Προτείνω να σα αφήσω εδώ ε, ένα αντίτυπο και στη γραμματεία ώστε να μπορέσετε να το ζητήσετε όσοι το θέλετε. Θα σας το διαθέσουμε χωρίς πρόβλημα. Υπάρχει όμως και μια έκθεση που έγινε το 2017 για την κατάσταση μέσα στην Ένωση. Εκεί περιγράφονται όλες οι χώρες και πρώτη και καλύτερη η Ελβετία που συνεχίζει να ε, φυλακίζει παιδιά 15 με 18 ετών σε κάποια από τα καντόνια. Δεν είναι και τέλεια, αν και όντως γίνονται πολλά πράγματα και στην Ελβετία. Καλά παραδείγματα. Έχουμε κάποια. Εμείς θα θέλαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης να συνεχίσουμε αυτήν την εξαιτία ώστε πραγματικά να φτάσουμε σε χώρες με βουλευτές, ώστε να μπορέσουμε να επισκεφθούμε τι γίνεται θετικό να έχουμε επαφή, το, επαφή ανάμεσα στις γραμματείες μας ώστε ίσως να ξεκινήσουμε τέτοιες επισκέψεις στο Ευρωκοινοβούλιο ας πούμε στο κέντρο Μπαρέκ στην Ελβετία να δείτε πώς με, ένα, με, ένα, με μια άλλη νοοτροπία μπορούμε να προχωρήσουμε. Να αναφέρω ποιες είναι εναλλακτικέ στην φυλάκιση, στην κράτηση και θα είμαι σύντομος. Τοποθέτηση σε δομές υποδοχής, οικογένειες υποδοχής, είναι κάτι το οποίο είναι αποτελεσματικό. Οι άνθρωποι είναι σωστοί και τα παιδιά έχουν πολύ καλή μεταχείριση, αντιμετώπιση. Δομές υποδοχής όπως ε, στο μπαρέκ, δηλαδή εστίες ε, ε, στέγασης. Αυτά κοστίζουν και πολύ λιγότερο από τη φυλάκιση και επιτρέπουν τον σεβασμό και την, την ανθρώπινη υποδοχή. Μπορούμε να έχουμε και δομές ε, ανοιχτές ή, ή μη ανοιχτές. Ε, στην Ελβετία υπάρχει ένα τέτοιο, ε, μια τέτοια δομή όπου τα παιδιά έρχονται και τα απασχολούμε. Μπορούν να έρθουν καθημερινά. Ε, επίσης ένα σύστημα όπου θα πρέπει να χτυπάνε κάρτα, ας πούμε, σε κάποιο δημόσιο ε, χτίριο. Ε, επίσης μπορούμε να κάνουμε, να μπορούν να μένουν σε συγκεκριμένα σπίτια, αλλά όπου δεν θα μπορούν να φύγουν από εκεί. Επίσης δομές με, ατομική προσέγγιση, ώστε να χαράζουμε ένα μέλλον για το παιδί. Να μην αισθάνεται μόνο του, να αισθάνεται ότι είναι ε, πλαισιωμένο. Με ατομική επίσης παρακολούθηση, με κοινωνικούς λειτουργούς που δημιουργούν μια επαφή με το παιδί, ε, αυτό του προστάτη, όπου οικοδομείται εμπιστοσύνη, μια σύνδεση με τις αρχές βέβαια και το παιδί καταλαβαίνει, αισθάνεται όπως κάποιος το κατανοεί και δεν θα φύγει, δεν θα προσπαθήσει να ε, το σκάσει. Μετά για τα, άτομα που έχουν κάποια χρήματα να μπορούν να δίνουν ας πούμε κάποια εγγύηση και το τελευταίο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ας πούμε μια ηλεκτρονική παρακολούθηση με ένα βραχιόλι ηλεκτρονικό. Εντάξει, ήδη αυτό είναι πιο οριακό αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι φυλάκιση και όλες αυτές οι μέθοδοι κοστίζουν πολύ λιγότερο από τη φυλάκιση και δημιουργούν πολύ λιγότερα προβλήματα στα παιδιά. Κάποιε φορές έχουμε εντύπωση ότι μπαίνουν στη φυλακή τα παιδιά πολύ μικρή ηλικία επειδή τα, οι γονεί τους κρατώνται. Πάντως ε, ε, θα πρέπει να ξέρετε ότι ένα παιδί όταν βλέπει τους, τους γονείς του να υποφέρουν, να είναι αδύναμοι και να είναι μέσα στο στρες και στην αγωνία, ε, μπορεί αυτό να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις γιατί τα παιδιά είναι σαν τα σφουγγάρια. Αυτό που, το χειρότερο που έχω δει είναι στο, στα τόπε, στο καταβλισμό Ρέσκε, στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας, με, από την πλευρά της Ουγγαρίας, όπου είδα πολλά α, σειρματοπλέγματα, πολλά παιδιά φυλακισμένα, δίχρονα, που παίζανε μπάλα με τους γονείς τους πίσω από ψηλά, ψηλούς φράχτες, παιδιά, με, ας πούμε είδα ένα παιδί 15 χρονών που είχε ε, μόνο το αυτοτραυματιστή είχε κοπεί, είχε ε, αυτά είναι στην δική μας Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πραγματικά είναι κάτι το α, απαράδεκτο. Ε, ε, σας ε, πιέζει ο χρόνος, θα σταματήσω λοιπόν εδώ, αλλά πραγματικά και γνή σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φριντές και εμείς ε, και σας συγχαίρομαι και αφού φτάσαμε σε αυτό, στο τέλος της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Θέλω να ευχαριστήσω τους ε, διερμηνείς για τα επιπλέον ε, λεπτά. Σας ευχαριστώ όλους που επιβιώσατε ε, σε αυτή την τελευταία μας συνεδρίαση και σας εύχομαι καλή ανάπαυση στη διάρκεια των διακοπών γιατί μας περιμένει πολλή δουλειά μετά. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Merci.